Um, Καλημέρα συνάδελφοι, ξεκινήσουμε εδώ στη γεμάτη αυτή η αίθουσα. Τόσοι πολλοί ενδιαφερόμενοι, πόσοι. Δύο, τρει, τρει βουλευτέ. Θαυμάσια. Ε, θα αποφασίσουμε και γρήγορα. Ίσως να κάνουμε τις ψηφοφορίες τώρα. Είναι κάποιο κατά? Όχι, εντάξει, εντάξει. Αστείευομαι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το σημείο 7. Πράσινη βίβλος. Δεν είναι εδώ. Α, εδώ είναι, εντάξει. Α, με, συγγνώμη, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ορίστε. Τρεις συν μία. Η Ματίας είναι εδώ και θα μας πληροφορήσει. Παρακαλώ λοιπόν, ξεκινήστε. Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κοιτάξτε, για μένα καλή είναι η ιδέα να αρχίσουμε με τις ψηφοφορίες. Έτσι θα είχαμε το 1 τέταρτο των ψήφων στην Επιτροπή. Δεν γίνονται όμως αυτά τα πράγματα, οπότε θα συνεχίσουμε με αυτό που είχαμε προγραμματίσει για σήμερα, δηλαδή συζήτηση για το στρατηγικό πλαίσιο, το κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την καινοτομία και την έρευνα και τη χρηματοδότηση του τομέα αυτού. Είναι μια πρώτη συζήτηση, μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Θα ήθελα να σας πω εξ αρχής ότι τα θέματα που θα θέσω είναι εξαιρετικά γενικά προς το παρόν. Κατόπιν σύν χρόνο θα εμβαθύνω αυτά τα ζητήματα σε συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές και τα λοιπά μέλη των ε, άλλων πολιτικών ομάδων. Ε, γνωρίζουμε όλοι ότι μας πιέζει το χρονοδιάγραμμα, είναι επίγον ε, το ζήτημα. Πρέπει να εκπονήσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου για αυτό το θέμα το ταχύτερο δυνατόν. Ε, γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να προσδώσουμε τη δέουσα σημασία στο ζήτημα και να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια παρά την πίεση του χρόνου. Τούτου θα αρχίσω την παρουσίασή μου λέγοντας ότι αυτό το κοινό στρατηγικό πλαίσιο ε, ενέχει πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και θα πρέπει να τα εξετάσουμε με προσοχή, με σαφή προσανατολισμό, κυρίως για το μέλλον της ε, ευρωπαϊκής έρευνας, ε, δοθήσεις της σημασίας της. Νομίζω κανείς δεν θα το αμφισβητήσει αυτό. Τώρα, ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές κάποιες από τις βασικές αρχές ε, που εξέθεσε στην Πράσινη Βίβλο της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι οι βασικές αυτές προκλήσεις, οι βασικές αυτές αρχές απορρέουν από προηγούμενες αξιολογήσεις των διαδοχικών προγραμμάτων πλαίσιο και ε, μέσων που είχαμε στον τομέα αυτό. Οι εξή αρχέ είναι ιδιαίτερε σημαντικέ. Πρώτον, να διευκρινίσουμε του στόχου. Δεύτερον, να μειώσουμε την περιπλοκότητα τη διαδικασία, να ενισχύσουμε την προσθέμενη αξία τη ευρωπαϊκή έρευνα στην παγκόσμια κλίμακα να απλουστεύσουμε την συμμετοχή. Έχουμε επιμακρύν συζητήσει αυτό το θέμα σε διάφορες συνεδριάσεις της Επιτροπής μας. Πέμπτον, ε, θα πρέπει να ενισχύσουμε τη συμμετοχή στα ερευνητικά προγράμματα που ήδη τρέχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ερευνητικά προγράμματα και προγράμματα καινοτομίας. Έκτον, να τονίσουμε πόση σημασία έχει η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών ε, που απορρέουν από τις δράσεις Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, στον τομέα της έρευνας. Αυτές οι έξι διαστάσεις του ζητήματος είναι οι πλέον σημαντικές και θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της πράσινης βίβλου. Υπάρχουν βέβαια και άλλες αρχές αλλά θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ανησυχία μου, διότι γνωρίζουμε την περιπλοκότητα του συστήματος, ε, τη διαρκή εναλλαγή των μέσων χρηματοδότησης που δυσχεραίνει την ε, ε, υλοποίηση, την περάτωση του κοινού ευρωπαϊκού χώρου έρευνας. Επανειλημμένα το έχουμε αναφέρει αυτό στις συζητήσεις της Επιτροπής μας, αλλά σε σχέση με αυτό θα έλεγα ότι θα πρέπει να στραφούμε προς τις βασικές αρχές του κοινού στρατηγικού πλαισίου για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή θα πρέπει να μειώσουμε τις επικαλύψεις και τον κατακαιρματισμό των προσπαθειών. Αντιλαμβάνομαι πλήρω του λόγου για του οποίου τίθενται αυτέ οι αρχέ μέσα στην πράσινη βίβλο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πλην όμω καταλαβαίνουμε επίση ότι όλοι θα πρέπει να συμβάλλουμε ώστε να μειωθούν οι επικαλύψει και ο κατακαιρματισμό. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τελείως βέβαια τον κατακαιρματισμό, ε, διότι Γνωρίζουμε ότι η αποτελεσματικότητα των ε, δράσεων συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, είναι συνάρτηση αυτών των αρχών που συνιστούν τις προτεραιότητες για μας, τόσο ώστε να κατοχυρώσουμε την επιστημονική συνεργασία και την αριστεία σε όλα τα ερευνητικά ιδρύματα της Ένωσης. Ε, θα έπρεπε σε τοπικό επίπεδο να ενισχύσουμε τις διαδικασίες ε, ενίσχυσης ε, των κοινοτόμων ερευνητικών μονάδων, ιδιαίτερα διαφοροποιημένων, κυρίως όταν θέλουμε να υλοποιήσουμε ταυτόχρονα τον στόχο της συνοχής για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Θα πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, προκλήσεις ε, με εξορθολογισμένο τρόπο, ούτως ώστε ε, να μην επιτύχουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση, βέβαια καλοπροαίρετα, διότι αυτό σημαίνει ότι τα ερευνητικά ιδρύματα θα έχουν λιγότερα μέσα στη διάθεσή τους, κυρίως σε κράτη-μέλη που για διάφορους λόγους, λόγω διαφόρων συγκυριών, ε, βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση. Ε, η επιστημονική αριστεία θα πρέπει λοιπόν να χρηματοδοτείται μέσω των εφιστάμενων ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Ε, θα ήθελα επίσης να κάνω ένα σχόλιο για την τωρινή ε, κατάσταση ύφεση, κρίσης, οικονομικής ε, και κοινωνικής βαθύτατης κρίσης ανά την, σε όλη την Ευρώπη. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι αυτό είναι πρόσκομα ε, που εμποδίζει την πρόοδο στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι η κρίση είναι μια ευκαιρία ε, για να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας ε, και να ανταποκριθούμε, να αντεπεξέλθουμε στην κρίση. Βεβαίως υπάρχει και μια αντίφαση και καλό θα ήταν να τη σχολιάσω εν παρόδο. Έχουμε ε, περισσότερες δημόσιες επενδύσεις για την έρευνα στην Ευρώπη σε σχέση με τη ΣΥΠΑ, πλην όμως τα αποτελέσματα και η αναγνώριση των αποτελεσμάτων υστερεί ε, έχουμε λιγότερες επενδύσεις ταυτόχρονα στον τομέα της ανώτερης εκπαίδευσης σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Αυτό το σχόλιο ε, έχει ιδιαίτερη σημασία και θα ήθελα να ε, τοποθετήσω αυτό το θέμα στον πυρήνα της ε, συζήτησής μας, διότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την εξής κατάσταση. Η έλλειψη εξαιρετικά ε, εξειδικευμένου προσωπικού στα ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα θα μπορούσε να στραγγαλίσει την ίδια την πρόοδο και την ε, εγκαθίδρυση την ίδια του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Οπότε θα πρέπει να αναρωτηθούμε ε, σε ποιο βαθμό έχουμε επαρκείς επενδύσεις στον τομέα της δημόσιας ανώτερης εκπαίδευσης και στον τομέα της ανάπτυξης και της έρευνας. Μήπως θα έπρεπε να ενισχύσουμε τα μέσα στους τομείς αυτούς. Εγώ πιστεύω πως ναι, με τρόπο ώστε να κατοχυρώσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα έχουν όλα τα απαιτούμενα κίνητρα ώστε να ενισχύσουν τις δημόσιες δαπάνες τους στον τομέα της ανώτερης παιδείας για να εξειδικευτούν ε, οι επιστήμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να στελεχώσουν τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. Ε, προς το παρόν όλα αυτά εξαρτώνται από την περιστασιακή εργασία πολλών επιστημόνων σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει και νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη πέραν από όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στην πράσινη βίβλιο της Επιτροπής. Ένα άλλο σχόλιο τώρα. Λαμβάνοντας υπόψη την ε, κατάσταση ε, που βιώνουμε, δηλαδή της λιτότητας, ε, της βαθιάς περιστολής των δημοσίων δαπανών, της βαθύτατης ύφεσης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, Θεωρώ ότι είναι μάλλον αυτονόητο ότι πρέπει να διατηρηθούν τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων διότι συνιστούν πυλώνα στις προσπάθειές μας για να αντιμετωπίσουμε αυτή την περιστολή των δημοσίων δαπανών και να δημιουργήσουμε μια Ευρώπη που θα αριστεύει και στον τομέα της καινοτομίας και έρευνας. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προβλέψουμε κίνητρα για τις περιφέρειες συνοχής ε, θα πρέπει αυτό να αποτελέσει έναν από τους φιλόδοξους στόχους της ευρωπαϊκής ερευνητικής πολιτικής και πολιτικής κοινοτομίας. Άλλες τρεις παρατηρήσεις ε, θα κάνω, διότι προφανέστατα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων σε αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Τέλος πάντων θα ήθελα να κάνω παρόλα αυτά άλλες τρεις παρατηρήσεις. Πρώτον, θα πρέπει αναμφισβήτητα, πέραν κάθε αμφιβολίας, να διευκρινίσουμε τους στόχους των επιμέρους ερευνητικών αναπτυξιακών προγραμμάτων ε, που χρηματοδοτούνται από τον περιπλογισμό της Ένωσης. Οπωσδήποτε θα πρέπει να προβούμε άμεσα στη διευκρίνηση των στόχων, κυρίως μέσα από τα μέτρα που ήδη παρουσιάστηκαν εν ώψη της απλούστευσης των διαφόρων ερευνητικών προγραμμάτων αναπτυξιακών προγραμμάτων και προγραμμάτων καινοτομία. Δεύτερη ε, παρατήρηση. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε τους λόγους για τους ε, οποίους παρουσιάζεται ως αδύρυτη ανάγκη να μεταφράσουμε τις επιστημονικές γνώσεις και ιδέες σε συγκεκριμένα προϊόντα και σε νέες υπηρεσίες εγώ θεωρώ ότι θα ε, οφείλουμε να υιοθετήσουμε μια ευρύτερη προσέγγιση, δηλαδή μια ευρύτερη αντίληψη του τι εννοούμε λέγοντας ε, ε, προϊόντα και υπηρεσίες, τι εννοούμε λέγοντας καινοτομία, κυρίως δοθήσεις της κρίσης που βιώνουμε. Και υπάρχει και κάτι που αναφέρεται, ελπίζω όχι εσκεμένα, μέσα στην ε, πράσινη βίβλο, γιατί ε, τονίζεται το βάρος ε, των προϊόντων και των υπηρεσιών, αλλά δεν αναφέρουμε πουθενά ότι οι επιστημονικές γνώσεις είναι δημόσιο αγαθό. Άρα, οι γνώσεις αυτές θα πρέπει να είναι προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπό αυτήν την έννοια, θεωρώ ότι η ενίσχυση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας ε, σημαίνει επίρρωσή σε παγκόσμιο επίπεδο, σε σύγκριση με όλες τις υπόλοιπε δυνάμει στην παγκόσμια σκηνή. Τέλος και θα κλείσω. Έχουμε συζητήσει διάφορα έγγραφα που σχετίζονται με το σημερινό θέμα με στόχο να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ε, μίζωνες κοινωνικές ε, προκλήσεις ε, που αντιμετωπίζει η Ένωση. Ε, δυστυχώς αυτό το έγγραφο δεν ε, πραγματεύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το θέμα και θα ήθελα με τη βοήθεια των συναδέλφων να συνδυάσουμε τις τεχνολογικές προκλήσεις με τις κοινωνικές προκλήσεις διότι υπάρχουν και είναι πολλές και δύσκολα μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε και γι' αυτό το λόγο και πάλι όπως σας έχω πει στο παρελθόν θα επαναλάβω ότι ε, δεν μπορούμε να ξεχνάμε τις ανθρωπιστικές επιστήμες που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ε, κοινωνικές ε, προκλήσεις. Ε? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αυξηθεί η χρηματοδότηση βεβαίως της επιστημονικής επιτροπής, το πρόγραμμα Marie Curie και όχι μόνο αλλά πέρα από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας ε, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε και τις ε, κοινωνικές ε, προκλήσεις διότι μην ξεχνάμε ότι δεν γνωρίζουμε καν όλα τα κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της Ένωσης και ξέρετε ότι σε αυτό έγκυται εν μέρη και η προστιθέμενη αξία της προσπάθειας που θα κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. ευχαριστώ. Οπότε σας ευχαριστώ και θα δώσω τον λόγο στους και Πρώτα απ' όλα λοιπόν η κυρία Χέρτσογκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως ο κύριος Χέκμαρκ είναι η μεγάλη, ανήκει στην μεγαλύτερη ομάδα. Ε, εγώ τον κατάλογο διαβάζω. Αν, εάν δεν θέλετε, ο κύριος Έλερ, ο επόμενος. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Ματίας. Δεν είμαι πολύ καιρό στο Κοινοβούλιο, αλλά πρώτη φορά άκουσα πως ε, η συγγήτρια ενδιαφέρεται για το τι κάνουν οι άλλοι. Δεν ξέρω τώρα το εννοεί στα αλήθεια ή αν είναι κάποια ευγένεια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το ασυνήθιστο και πολύ φιλικό. Δύο παρατηρήσεις πρώτα απ' όλα. Το θέμα του πώς θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα πλαίσιο 8 είναι κατά βάση το ερώτημα του εάν θα παραμείνει κάτι από τη, από τη στρατηγική της Λισαβόνας. Βλέπουμε στις εκθέσεις όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα και τους υψηλούς στόχους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο το να μπορέσουμε να σταθούμε στο ίδιο ύψος με την Αμερική και τις εξελίξεις στην Ασία που ήταν ο στόχος ε, ότι έχει αποτύχει οπότε όσον αφορά το πρόγραμμα πλαίσιο 8 θα πρέπει να έχουμε πιθανότατα μία μείωση. Και βέβαια στο πλαίσιο, πρόγραμμα πλαίσιο 8 έχει τόσο μεγάλη σημασία γιατί το θέμα είναι τι έχει απομείνει από του όχου τη Λισαβόνα και το εάν είμαστε στη θέση πλέον εδώ μέσα να διαμορφώσουμε ένα δυναμικό, οικονομικό ε, και ισχυρό στόχο όσον αφορά τις προοπτικές. Εάν παραμείνουμε τώρα τα πλαίσια του προγράμματος 7, τότε δεν θα μείνουμε απλά στο status quo, αλλά θα παραμείνουμε σε ένα αραβούργημα, δηλαδή μια φιλική χειρονομία προς την ευρωπαϊκή ιδέα, αλλά δεν θα έχει κάποια, κάποιο πραγματικό αντίκρισμα. Οπότε είναι ε, το ζήτημα εδώ πέρα κάτι το οποίο σχετίζεται με το εάν πραγματικά θέλουμε μια Ευρώπη ε, κοινή και πάει παραπέρα από το ζήτημα απλά ενός αριθμού στο συνολικό προπολογισμό ή της πολιτικής της έρευνας. Οπότε είναι σαφείς οι συνθήκες. Πρέπει λοιπόν ως Κοινοβούλιο να σκεφτούμε το εάν θα βρούμε μια κοινή στάση και αυτό θα αποτελέσει τη μοναδική ευκαιρία για να επηρεάσουμε την συγκρατημένη να θέση της ε, Κομισιόν και την πολύ επιφυλακτική θέση του Συμβουλίου για να προωθήσουμε αυτό το πρόγραμμα για να αποκτήσει και μία ουσία. Γι' αυτό θεωρώ πως είναι σημαντικό εκ των προτέρων να ξεκαθαρίσουμε ποιο είναι το θέμα. Ε, εάν τους στόχους που έχουμε ορίσει οι ίδιοι θέλουμε να τους επιτύχουμε πρέπει να έχουμε διπλασιασμό του προϋπολογισμού. Μόνο έτσι είμαστε στο ίδιο επίπεδο με τις εξελίξεις στην Αμερική και την Ασία. δεύτερον, έχουμε μια σύγκρουση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Το είχαμε λύσει αυτό τότε από κοινού στο Κοινοβούλιο με της ε, διαπραγματεύσεις και είναι η σύγκρουση μεταξύ των νέων ας πούμε χωρών και των παλαιών μεταξύ των μεγάλων και των μικρών κρατών μελών. Ε, εν πάση περιπτώσει έχουμε δεσμευτεί για την αριστεία. Την αριστεία βασικό κριτήριο του προγράμματος πλαισίου αλλά πρέπει βεβαίως να πούμε πως ε, το αποτέλεσμα του εβδόμου προγράμματος ε, πλαισίου σημαίνει πως ε, υπήρχαν κρατημέλη τα οποία δεν μπορούσαν να λάβουν μέρος γιατί ακόμα οι δομές τους ήταν υποδιαμόρφωση και βεβαίως σε ορισμένα σημεία είναι αρκετά καλές αλλά δεν είχαν φτάσει στο επίπεδο το οποίο θα θέλαμε σε αυτά τα πράγματα στην Ευρώπη. Και βλέπουμε πως ε, από τη μία βεβαίως θα πρέπει οι νέες χώρες ε, να έχουν ε, ένα συμφέρον να συμμετέχουν περισσότερο στο πρόγραμμα και βεβαίως αυτό σημαίνει πως αυτό το απόλυτο κριτήριο της αριστείας αμφισβητήθηκε ως έναν βαθμό και από την άλλη υπάρχουν κράτη-μέλη που λένε πως εάν είναι να αμφισβητούμε το κριτήριο της αριστείας τότε δεν μας ενδιαφέρει εμάς να στηρίξουμε αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα και θα τα κάνουμε με τα εθνικά προγράμματα. Πρέπει να μιλήσουμε ανοιχτά για αυτό το θέμα και να βρούμε νωρί έναν συμβιβασμό, αλλιώς θα διχαστούμε, θα διχαστεί το Συμβούλιο και δεν θα έχουμε ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη για το πρόγραμμα 8. Οπότε, θα πρέπει να πούμε πως το κριτήριο είναι η αριστεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τον ανταγωνισμό παγκοσμίω, αλλά από την άλλη αναζητούμε μία λύση για το πως θα μπορέσουμε να συμβάσουμε τα διαφορετικά συμφέροντα. Αυτό το οποίο είπαμε δηλαδή ως τίτλο μία σκάλα η οποία θα οδηγεί προς την αριστεία. για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες ε, δομές οι οποίες θα οδηγήσουν κάποια κράτη-μέλη προς ε, την ε, αριστεία. Εάν επιτύχουμε αυτόν τον συμβιβασμό και έχουμε ισχυρή θέση του Κοινοβουλίου, θα είναι οπωσδήποτε θετική εξέλιξη. Αλλιώς βεβαίως θα είναι και εξαστερημένη και η θέση του Κοινοβουλίου. Το τρίτο μεγάλο θέμα είναι το θέμα το οποίο συζητιέται, σε ποιο ε, βαθμό ε, το πρόγραμμα αυτό πλαίσιο εξυπηρετεί την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και είναι σαφές πως πρέπει να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ της απαραίτητης θεμελιώδους βασικής έρευνας που είναι βεβαίως ε, το ισχυρό σημείο της έρευνας στην Ευρώπη και από την άλλη να δούμε πώς θα ε, έχουμε εφαρμοσμένη έρευνα, εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας, καινοτομία, πώς θα μεταφραστούν όλα αυτά σε συγκεκριμένα προϊόντα, σε οικονομική ανάπτυξη. Οπότε έχουμε το ζήτημα που σχετίζεται με το πρόγραμμα 8 για το ποια μέσα θα ενσωματώσουμε το CIP, παραδείγματος χάρη, θα ενσωματωθεί στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο ή το πρόγραμμα πλαίσιο είναι ξεκάθαρα πρόγραμμα καθαρής έρευνας ή είναι έρευνας και ανάπτυξης. Θα μπορέσει να συνδεθεί δηλαδή με το CIP έτσι ώστε με συγκεκριμένα μέσα να χρησιμοποιηθούν αυτές οι τεχνολογίες στις χώρες. Είναι ένα θεμελιώδες στρατηγικό ερώτημα, γι' αυτό χαιρετίζω εγώ το ότι στην Κομισιόν, η Κομισιόν παρά το ότι είναι ασαφής στην Πράσινη Βίβλο θέτει στο προσκήνιο την καινοτομία για να υπάρξει και ανάπτυξη στην Ευρώπη. Τελευταίο θέμα, μάλλον τα δύο τελευταία, είναι αφενός η διεθνής συνεργασία. Μιλάμε για διεθνή συνεργασία, αλλά ο απολογισμός του προγράμματος 7 είναι πολύ πενιχρός. Δηλαδή, για πολλές χώρες, ερευνητικά ιδρύματα και στην Ασία και στη Βόρεια Αφρική. Ε, δεν είναι ελκυστικό το πρόγραμμα γιατί κινούνται πολύ αργά οι διαδικασίες, γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις στην ε, Ασία στον τομέα της πληροφορικής που είναι πολύ δυναμικές και δεν βρίσκουν ε, κάποιον εταίρο για επιστημονικά έργα στην Ευρώπη γιατί χρειάζονται 1,5-2 χρόνια για να ληφθεί μια απόφαση δεν είναι ανταγωνιστικό εντό αγωγικών αυτό σε διεθνέ επίπεδο. Δηλαδή πρέπει να δούμε το θέμα τη διεθνού συνεργασία πολύ περισσότερο και να σκεφτούμε ποιε διαρθρωτικές αλλαγές πρέπει να γίνουν για να είναι πιο ελκυστικές οι μορφές αυτές έγκρισης σε διεθνές επίπεδο. Το τελευταίο θέμα το οποίο δεν αναφέρεται στο βράσινο βίβλιο αφορά την χρηματοδότηση των μεγάλων ευρωπαϊκών έργων. εμέσως χρηματοδοτούμε πολλά μεγάλα ευρωπαϊκά έργα όπως το GNS ε, Ήτρε και τον Γαλιλαίο και μπορούμε να προβλέψουμε πως δεν θα μπορεί να γίνει αυτό πλέον μέσω του κλασικού προπολογισμού. Το, να σας υπενθυμίσω τι έγινε με την προσπάθεια συμβιβασμού για το Ίτερ το Δεκέμβριο γιατί προσπαθήσαμε να βρούμε κονδύλια που είχαν απομείνει στη Γεωργία, στον πυλώνα 2 για να πάνε στη χρηματοδότηση ενός μεγάλου ευρωπαϊκού έργου. Δεν τα καταφέραμε. Και είναι σαφές πως και με το τρέχον πρόγραμμα 8 δεν θα καταφέρουμε να χρηματοδοτήσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις είτε GNS και Γαλλιό. Χρειαζόμαστε μια ξεχωριστή γραμμή του προπολογισμού για τη χρηματοδότηση μεγάλων ευρωπαϊκών έργων. Από ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει δεν θα μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε αυτά τα έργα. Μπορούσε να γίνει αυτό στην αρχή, αλλά σε βάθος χρόνου θα πρέπει να υπάρχει ένας ξεχωριστός ε, τίτλος στον προπολογισμό. Και τελευταίο, γιατί τον τονίζουν όλοι οι συνάδελφοι και εγώ πάντα στις ομιλίες που κάνουμε και πάντα λέμε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως εποδό. Ε, κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσουμε για κάποια ουσία σε αυτό το πράγμα. Είτε είμαστε πραγματικά διατεθειμένοι να πούμε πως θα έχουμε πραγματικά απλοποιημένες διαδικασίες σε ορισμένους τομείς και θα τις αποδεχτούμε γιατί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν μπορούν να ενσωματωθούν στο πλαίσιο πολυετών προγραμμάτων ή να πούμε πως είναι απλά κάτι, μια υποδόση. έτσι κάτι που το λέμε για να το λέμε. Γιατί βλέπετε σε πέντε διαδοχικά προγράμματα μειώνεται το ποσοστό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κάποια στιγμή θα μας πούν πως ε, μόνο λόγια λέμε και στην πράξη δεν κάνουμε τίποτα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να έχουμε τομεακές προσεγγίσεις για τις, ε, μικρομε... για ε, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Να έχουμε μια τομεακή προσέγγιση γιατί δεν μπορεί να έχουμε από ένα ελληνικό περίπτερο μέχρι μια σουηδική επιχείρηση την ίδια αντιμετώπιση. Και να πούμε πως ε, ισχύει για όλους τους κλάδους ε, της βιομηχανίας. Αλλά όταν μιλάμε για μικρομεσαία επιχείρηση ε, π.χ. στον τομέα της πληροφορικής έχουμε κάνει πολύ στενό τον ορισμό γιατί θα μπορούσαμε να καλύψουμε πολύ περισσότερα από το πλαίσιο το οποίο υπάρχει τώρα. Οπότε χρειάζονται εδώ πέρα πιο έξυπνες λύσεις τομεακές, όπως είπα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Έχω ακόμη έξι συναδέλφους, κομισιόν και εισηγήτρια και 10 η ώρα ψηφίζουμε. Οπότε παρακαλώ να είστε σύντομοι ή οι τελευταίοι δεν θα μιλήσουν διαφορετικά. Λοιπόν, η κυρία Χέρτσογκ κατόπιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ήθελα να τηρήσω το πρωτόκολλο να μιλήσουν οι, οι εκπρόσωποι των μεγαλύτερων κομμάτων. Να είμαστε όμω και αποτελεσματικοί. Γιατί, οπότε να μην επαναλάβω αυτά που είπε ο εισηγητή από το ΕΛΚ. Για να δούμε. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θέλει να προχωρήσουμε με επιτυχία προς την επίτευξη των στόχων του 2020 και αυτό καλύπτει και την καινοτομία και την έρευνα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. Πρόκειται για μια μεγάλη πρόκληση και η διαδρομή να αρχίσει σήμερα. Όλοι συμφωνούμε επίσης ότι θα ε, πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε δαπάνε, θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή κρατών μελών και τη Ένωση, όμω, μέχρι σήμερα τα έχουν πάει τόσο καλά. Και το θέμα είναι μήπως οι Υπουργοί Οικονομικών άλλα λένε στην ε, Ένωση και άλλα λένε στις κυβερνήσεις και εν πάση η δική τους γνώμη περνάει και όχι η γνώμη άλλων Υπουργών. Συμφωνήσαμε όμως για την καινοτομία. Συμφωνήσαμε και να έχουμε λύσεις διαφοροποιημένες. Όπως είπε και αποτέλεσμα να καλύψουν και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Άρα, το πρόβλημα ποιο είναι. Θα πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι ότι έχει αλλάξει τελείως το τοπίο όσον αφορά την καινοτομία. Καινοτομία και έρευνα δεν αφορά μόνο τι εταιρείε τεχνολογία αιχμή. Αφορά και την κοινωνική καινοτομία, αφορά και το δημόσιο τομέα. Και οπότε θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι εάν δεν διπλασιάσουμε, τριπλασιάσουμε του πόρου που διατίθενται, τότε ας κρατήσουμε την πρεκοδότηση του 7ου προγράμματος πλαισίου. Αλλιώς συρρυκνωνόμαστε. Γιατί αν ανεβαίνει ο πύχης και μένουν ίδια τα χρήματα είναι σαν να μειώνονται. Άρα θα πρέπει να αυξηθεί το ποσό και άρα να είμαστε ενωμένοι και να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερη προκοδότηση από όσο ισχύει σήμερα και νομίζω πάντως ότι η δική μας Επιτροπή όντως είναι ενωμένη σε αυτό. Τώρα, Υπάρχει εδώ ένα πρόβλημα. Το πέμπτο κεφάλαιο. Εκεί που λέμε για τις διοικητικές δαπάνες, μια που τα περισσότερα αφορούν αυτές τις διοικητικές δαπάνες. Αλλιώς θα πρέπει να συνδυάσουμε τους πόρους που θα έχουν στη θέση μας. Να δούμε επομένω το κάθε κονδύλιο χωριστά για να δούμε αν μπορούμε να καλύψουμε όλους τους επιμέρους στόχους μας. Επίσης, θα πρέπει να γίνει αναθεώρηση της πολιτικής κοινοτομίας, όπως επίσης και το ευρωπαϊκό ε, την Ευρωπαϊκή για την Καινοτομία. Για να προσθέσουμε γιατί προβλέπεται με τη συγχρηματοδότηση απολύτω τα κράτη-μέλη, τα κονδύλια του τα παίρνουν πίσω και θεωρούν ότι θα του καλύψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ θέλουμε τα κράτη-μέλη να πετύχουν αποτελέσματα. Δεν πρόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση να αφαιρθεί σαν φιλανθρωπικό ίδρυμα και να χαρίζει αυτά στα κράτη-μέλη. Για τα προγράμματα που έχουμε τώρα, το Γαλιλαίο και τα άλλα, να πάμε για την αύξηση το 3% του ΑΕΠ και θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη μας κατά των Υπουργών Οικονομικών. Αλλιώ θα χάσουμε αξιοπιστία γιατί έχουμε κάποιε υποσχέσει από μια μεριά, αλλά από την άλλη μεριά χρειάζονται και τα μέσα για να υλοποιηθούν οι υποσχέσει. Δεν θα πρέπει το Κοινοβούλιο να συμμετάσχει σε κάποιο τέτοιου παιχνιδάκια και ξεγέλασμα του κόσμου. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Um, I would uh, like to state... Uh, Κατά τη γνώμη μου, να σας πω ποια θα πρέπει να τα βασικά όσον αφορά την επόμενη γενιά προγραμμάτων για καινοτομία. Να δούμε τι θα γίνει στον πρωτιστική και Δαπάνη, Θα πρέπει επίση να έχουμε επίδειξη, αξιολόγηση αποτελεσμάτων και καινοτομία. Όπως που ο κ. Χέλλερ, πρέπει να συνδυάσουμε την αριστεία αλλά και την κλίμακα της αριστείας να καλύψουμε. Όπως το είπε ο κύριος Σέλλερ και άλλοι συνάδελφοι θα πρέπει να διπλασιαστεί η πρικοδότηση για αυτά τα οποία θέλουμε. Και επίσης θα πρέπει να προχωρήσουμε σε λύσεις συνεργασίας. Να δούμε τι θα γίνει με το 8ο πρόγραμμα πλαίσιο για πληροφορική κλπ. Αλλά έχουμε πολιτική και βιομηχανία σαν άλλους πυλώνες στο πρόγραμμα πλαίσιο. Χρειάζεται να πετύχουμε ισόρροπες λύσεις όσον αφορά την έρευνα προσέγγιση από πάνω ή από κάτω ή από τη βάση από τη βάση το Συμβούλιο Έρευνα. Αυτό θα πρέπει να αφορά και το πρόγραμμα συνεργασία. Κάτι γνώμη μου. Το πρόγραμμα συνεργασία είναι στοιχείο πάρα πολύ σημαντικό του 7ου προγράμματο και να συνεχίσει να είναι και στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Θα μπορούσε βέβαια αυτό να γίνεται κείμενο συνεργασία, προσέγγιση από τη βάση προ την κορυφή. τελικά αυτοί που θα συμμετάσχουν θα ορίσουν ποιες αναδυόμενες τεχνολογίε θα χρησιμοποιηθούν για τους επιστημονικούς τομείς. Είπαμε να αλλάξουν οι κανόνες γιατί τα προγράμματα θα πρέπει να πιο προσβάσιμα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις άρα να επανασχεδιαστούν. Γιατί προς το παρόν οι επιλέξιμοι κυρίως είναι, δεν είναι οι ίδιες οι μημιές αλλά κυρίως κάποια ερευνητικά ιδρύματα. Άρα να δούμε με ποια συγκεκριμένα μέσα θα τους διευκολύνουμε. Και έρευνα και ανάπτυξη να αποδώσει καρπούς και σε επίπεδο αγοράς. Αυτό είναι ένα στόχο Θα πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο οι νέοι επιστήμονε θα μπορέσουν να συμμετάσχουν περισσότερο στα ερευνητικά προγράμματα και για βιομηχανία και για ερευνητικά ιδρύματα. Τελευταίο τώρα. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις ε, διατάξεις απλούστευσης που δεν ισχύουν για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Να δούμε κυρίως τι θα γίνει με τον δημοσιονομικό οργανισμό. Παρακολουθούμε επομένως τι γίνεται με αυτές τις αποσυντικές διατάξεις και θα προσπαθήσω με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσω τον εισηγητή. Πρόεδρος. Χόκμαρκ. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και τον εισηγητή. Ε, είμαι στην ευτυχή θέση να συμφωνώ με όλους Πολύ καλό αυτό. Αυτό δείχνει ότι έχουμε την κατεύθυνση που να ακολουθήσουμε μπροστά μας. Επίσης, να δούμε τι γίνεται με ε, ε, ε, το βασικό θέμα εδώ που είναι η απλούστευση. Απλούστευση και πάλι απλούστευση αυτό χρειάζεται. Και επομένως, με την απλούστευση όχι μόνο αντιμετωπίζουμε γραφειοκρατία, αλλά αποτελεί η δουλειά μας ε, πόλο έλξης αποκτά δυναμισμό. Να πετύχουμε αυτά που δεν πετύχαμε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Ακόμα έχουμε δουλειά μπροστά μας. οι μικρομεσαίες εταιρείε, όλοι όσοι συμμετέχουν στην καινοτομία, όλοι όσοι δίνουν δυναμισμό σε επιχειρήσεις να ελκυστούν. Επίσης, να δούμε τι γίνεται το επίπεδο χρηματοδότησης. Είπαμε ότι στόχος μας είναι να διπλασιάσουμε την πληροδότηση. Ο λόγος είναι απλός. Όλα ό,τι προβλέπετε μέχρι σήμερα έχει να κάνει με το ότι στην επιστημονική έρευνα κυριαρχεί η Αμερική και η Ευρώπη. Ρίχτε μια ματιά στο παρελθόν. Όλες οι προσπάθειες κατεβλήθησαν από Ευρωπαίους και Αμερικανούς. Αλλάζουν όμως τα πράγματα. Αλλάζουν γρήγορα και σήμερα. η Ινδία και Κίνα έχουν περισσότερους ερευνητές, μηχανικούς, ε, ε, επιστήμονες. Τα ξέρετε τα στατιστικά. Και αν εκτός μικροφώνου Πόσο, μόνο, 12, μόνο εκείνα έχει 12 εκατομμύρια. Να βλέπετε. Ευθυγραμμίζεται μαζί μου και η Γερμανία. Πάντα, πάντα έτσι. Να επομένω ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Το τελευταίο τώρα. Θα πρέπει η κινητικότητα των ερευνητών να αυξηθεί, Πρόεδρε. Να γιατί πήγανε καλά οι Αγγλοσάξονες και οι Αμερικανοί. Η κινητικότητα, η ευκολία προσβασιμότητα σε όλων αυτών των ανθρώπων στα ερευνητικά κέντρα. Και δεν πρόκειται μόνο για αναβάθμιση του προγράμματος ε, Μαρία Κιουρί. Γενικότερα θα πρέπει να δούμε πώς θα έχουμε ενίσχυση των πρωτοπόρων ερευνητικών ιδρυμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σοντή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τη Μαρίσα Ματίας ε, για την παρουσίαση που έκανε και η οποία καταδεικνύει το ανοιχτό της ε, πνεύμα ένα μεθοδολογικό πρόβλημα πρώτα απ' όλα. Λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να έχουμε τις προτάσεις μέχρι τον Ιούνιο 2011 για το μελλοντικό δημοσιονομικό πλαίσιο. Μα έχει καθυστερήσει για την αξιολόγηση του 7ου προγράμματος πλαίσιο και εμείς ε, έχουμε μπει μέσα σε μια κατεπίγουσα διαδικασία και θα κάνουμε καμιά βλακία γιατί όποιος βιάζεται σκοντάφτει. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια πολιτική συζήτηση για τα θέματα και έχω κάνει εξή εισήγηση. Αν μα πιέζει τόσο πολύ ο χρόνο, ε, τουλάχιστον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δεχτεί ε, να είναι πιο διαλλακτική. Δηλαδή, με το που λάβουμε το κείμενο μπορούμε να το τροποποιήσουμε αναλόγω από τι συγκυρίε. Για το 7ο πρόγραμμα δεν το κατάφερα, αλλά βάσει το άρθρο 138 τη συνθήκη επιτρέπεται αυτό ε, να προσαρμόζουμε το πλαίσιο δηλαδή στην ε, πραγματικότητα που ζούμε. Έχει αποτύχει η στρατηγική της Λισαβόνας, ε, βιώνουμε τη βαθύτατη κρίση από το 2008. Ε, είμαστε σε επισφαλή θέση και μας λένε δεν μπορείτε να τα κουμπίσετε το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Πολύ ωραία. Για το 8ο όμως ε, θα πρέπει να κάνουμε όλη μια εισήγηση για να είμαστε πιο διαλλακτικοί. Δηλαδή να γίνεται η αξιολόγηση και να δούμε αν χρειάζεται προσαρμογή το πρόγραμμα με τις νέες συνθήκες. Κάτι άλλο τώρα. Μέσα στην πράσινη βίβλο δεν αντιμετωπίζουμε σφαιρικά το πρόβλημα της έρευνας. Τι εννοώ λέγοντας σφαιρικά ε, πρέπει να καλύψουμε τις περιφέρειες, τα έθνη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τρία αυτά επίπεδα. Προτείνω το ελεγκτικό συνέδριο και τα 27 εθνικά ελεγκτικά συνέδρια να κάνουν έναν εξωτερικό έλεγχο στον τομέα της έρευνας για ολόκληρη τη γυραιά Ήπειρο. Δηλαδή, ωραία να διπλασιάσουμε τα κονδύλια, συμφωνώ. Αλλά πώς θα χρηματοδοτήσουμε θα πρέπει στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας να έχουμε όσο γνώμονα τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό των προσπαθειών μας. Δεν το καταφέρουμε αυτό αν δεν γίνει αξιολόγηση. Το Συμβουλίο της Ευρώπης επίσης έχει σημαντική συμβολή και αναφέρεται αυτό σε πολλά σημεία στην Πράσινη Βίβλο. Δηλαδή από κοινού και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δράσουν σε συνεργασία. Νομίζω ότι αυτό τι θα πρέπει να είναι η πρώτη στη αρχή στο 8ο πρόγραμμα πλαίσιο. Η κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ οργάνωσα ένα μικρό διάλογο με καθηγητές και διευθυντές Ινστιτούτων στην Πολωνία για να μου πούν πώς αξιολογούν τα βασικά προβλήματα του προγράμματος 7 και το τι περιμένουν. Κάποια ζητήματα αναφέρθηκαν ήδη. Εγώ ήμουν και καθηγήτρια και τα ξέρω και από μέσα. Κάποια προβλήματα αναφέρθηκαν, η υποδομή είναι κρίσιμη, πολλά από αυτά τα Ινστιτούτα δεν έχουν ε, αρκετά καλή υποδομή για να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους. Βεβαίω, τα ε, τυπικά ζητήματα είναι αφόρητα για τα Ινστιτούτα και τα Ιδρύματα εκείνα που δεν έχουν διοικητικές ικανότητες. Δηλαδή, ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους, ε, αλλά το ενδιαφέρον αυτό μειώνεται. Υπήρχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αρχή όταν είχαμε ενταχθεί στην Ένωση, τώρα μειώνεται. Νομίζω πως αυτό είναι πάρα πολύ κακό σημάδι και αυτό το ζήτημα του υπάρχοντος ε, και μεγάλου αναπτυσσόμενου κενού πρέπει να συζητηθεί περισσότερο. Επίσης αυτό το οποίο λέμε για τις ε, τυπικές απαιτήσει. έχουμε πρώτα απ' όλα τις απαιτήσει εκθέσεων, ενδιάμεσων συχνά η αξιολόγηση είναι τυπική και όχι αξιοκρατική ε, όσον αφορά δηλαδή τα αποτελέσματα. Οπότε αν γίνει ένα λάθος ε, μένει κάποιος εκτός και όλοι τρέμουν, μην κάνουν κανένα λάθος γιατί δεν θα λάβουν τα χρήματα. Αντί να σκέφτονται και να κάνουν κάτι δημιουργικό. Δεύτερον, που αναφέρθηκε, είναι πως η καινοτομία γίνεται αντιληπτή υποτεχνικούς και όχι κοινωνικούς όρους. Σε αυτές τις χώρες μιλάμε για κοινοτόμε μορφές εργασίας, ε, υπάρχουν πολλά κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα. Ε, και η ερμηνεία είναι πολύ στενή εδώ πέρα. Μετά, πρακτική χρήση. Γιατί και αυτό αποτελεί κριτήριο. Τι σημαίνει αυτό σε γενικές γραμμές λένε πως οι κοινωνικές επιστήμες οι οποίες ε, μπορούν επίσης να έχουν καινοτομία αντιμετωπίζονται με πολύ χειρότερο τρόπο. Τα έργα είναι πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλα. Κοιτάξτε, εγώ συμμετείχα σε τέτοια έργα. Δεν ξέρουμε ποιος συμμετέχει, ποιος κάνει τι και προστίθενται έτσι μικρά λιθαράκια σε μια μεγάλη πυραμίδα. Δεν είναι καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα αυτά. Κάποια από αυτά, ε, κάποιοι, με συγχωρείτε από συνομιλητές μου, είπαν πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια κοινή πολιτική, πολιτική συνοχής όσον αφορά την έρευνα. Δεν θέλω εγώ να ακολουθήσω και αυτή την ιδέα, απλά προτάθηκε. Ε, δεν θα σπαταλήσω όλο το χρόνο, σας ευχαριστώ. Η κυρία Φόρτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ αναμένω βέβαια συνεργασία με την εισηγήτρια και τους σκιώδεις εισηγητές. Να αναφέρθω σε κάποια σχόλια των συναδέλφων. Υπάρχει ισορροπία αυτή μεταξύ, που θα πρέπει να βρεθεί βεβαίω, μεταξύ αριστείας και ευρύτερη συμμετοχής. Είναι ένα θέμα στο οποίο θα πρέπει να δώσει έμφαση το Κοινοβούλιο. Για τη συμμετοχή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το έχω ξαναπεί. Η απλοποίηση είναι το βασικό εδώ πέρα για να λάβουν μέρος και πολλές χώρες και διαφορετικοί φορείς. Όσον αφορά τα αποτελέσματα και τον προσανατολισμό στα αποτελέσματα, ναι, όπου ε, απαιτείται αυτό, γιατί δεν πρέπει να μιλάμε και να ζητάμε γενικώ ε, αποτελέσματα. Νομίζω η Μαρία Καρβάγιο είπε η ε, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και αυτό το οποίο ακούστηκε μια σκάλα που θα οδηγεί προς την αριστεία και αυτό θα έπρεπε να το δούμε. Επίσης, το ότι δεν ε, είμαστε αρκετά γρήγοροι στις αποφάσεις χρηματοδότησης των έργων και σημαίνει πως οι λοιποί διεθνείς εταίροι δεν συμμετέχουν. Ναι, δεν είμαστε αρκετά γρήγοροι, αλλά γι' αυτό ακριβώς και οι ευρωπαϊκοί φορείς συχνά δεν συμμετέχουν. Ειδικά αν είναι σε ένα κλάδο που έχει ε, μικρό χρόνο μεταξύ έρευνας και διάθεσης στην αγορά, π.χ. στην υψηλή τεχνολογία κτλ. Όπου πρέπει το προϊόν να βγει γρήγορα σε μια ανταγωνιστική αγορά παγκόσμια όταν χρειάζεται πολύ χρόνος για να ληφθεί μια απόφαση, ε, αυτό γίνεται μετά μη ανταγωνιστικό σε μια παγκόσμια αγορά. Και όταν μιλάμε για τη συνεργασία με διεθνείς φορείς. Ναι, εντάξει, αντιλαμβάνομαι την ανάγκη, αλλά ε, να έχετε κατά νου πως το πρόγραμμα πλαίσιο είναι το μόνο έργο στο οποίο μπορούν να εμπλακούν ε, διεθνείς φορείς δεν υπάρχει αλλού τέτοιο σύστημα για άλλα μέρη του κόσμου. Όσον αφορά το σχόλιο τώρα περί μιας ε, γραμμής προπολογισμού, ειδικά για μεγάλα έργα, πράγματι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια για το πού βρίσκονται αυτά τα μεγάλα έργα και αναμένω τις ε, σχετικές συζητήσεις. Το σχόλιο για την έμφαση σε ενεργειακή ασφάλεια, εξοικονόμηση ενέργειας κτλ. Χρηματοδοτούνται πολλά τέτοια έργα, ναι είναι σημαντικά. Οπότε πρέπει να δώσουμε βάρος σε μεγάλες προκλήσεις, ε, ενεργειακή ασφάλεια, ασφάλεια τροφίμων και να έχουμε αποτελέσματα. Επίσης, οι τρει πυλώνες, η έννοια αυτή, δηλαδή επιστήμης, βιομηχανίας και πολιτικής, μπορεί να είναι χρήσιμη έννοια. Η απλοποίηση είναι το κλειδί, θα έλεγα, για να επιτύχουμε πολλούς από τους στόχους μας. Τα σχόλια που έγιναν σε μένα ε, είναι πως ε, θα πρέπει να είναι απλά τα μέσα και μου λένε μην, να μην εισαχθούν νέα μέσα. Βεβαίως ε, όταν οι δαπάνες πιέζονται πρέπει να φροντίσουμε να ξοδεύονται σωστά οι επενδύσεις μας ε, και βεβαίως ίσως το να, το να αυξήσουμε αυτή, την, το μέσο ίσως να είναι καλύτερο. Ευχαριστώ κύριο Τσουκαλά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σύντομα, αποδέχομαι τις εισηγήσεις του κυρίου Έλερ και της κυρίας Καρβάλιο και εστιάζομαι στο, σε δύο ζητήματα. Το ένα ζήτημα είναι το ζήτημα της αριστείας. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει η αριστεία ή αλλιώς η επιλεκτικότητα στη χορήγηση των πόρων οδηγούν σήμερα την έρευνα στην ανάδειξή της. Ξαναφέρνω το παράδειγμα. Η Κίνα έχει 120 όλα και όλα πανεπιστήμια που δίνουν διδακτορικά και η Αμερική 238. Πρέπει στην Ευρώπη να επιδοτήσουμε την αριστεία και να επιζητήσουμε την κλίμακα προς την αριστεία μέσω της συνεργασίας των διαρθρωτικών προγραμμάτων με τα προγράμματα πλαίσιο θα έβλεπα εκεί την ανάγκη οι χώρες που παίρνουν χρήματα από τα διαρθρωτικά ταμεία και τα διαθέτουν για την έρευνα να υφίστανται τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τα προγράμματα πλαίσιο με εξωτερική αξιολόγηση των έργων τους. Η χρηματοδότηση μεγάλων ερευνητικών έργων και ε, υποδομών στην Ευρώπη είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό Τέλος, τελειώνω με την παρατήρηση ότι εμείς δεν πρόκειται να υπαγορεύσουμε στην πραγματικότητα πώς να φερθεί. Ήδη τα διεθνή δίκτυα μεταξύ των επιστημόνων, οι καινούριε αναδυόμενες μεγάλες ερευνητικές και επιστημονικές δυνάμεις. Το γεγονός που ανέφερε ο κύριος Λάγκεν ότι η Κίνα έχει 12 εκατομμύρια επιστήμονες πρέπει να προσθεθεί ότι η Κίνα βγάζει και 1,5 εκατομμύριο επιστήμονες το χρόνο και η Ινδία βγάζει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Η Αμερική από το 1 εκατομμύριο που δαπανάται για την έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο πληρώνει τα 400 δισεκατομμύρια, η Κίνα πληρώνει τα 100 δισεκατομμύρια και αυτά είναι μεγέθη τα οποία πρέπει να ξέρουμε. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός που ελέγχθη ως προς την έρευνα και την τεχνολογία για μένα είναι νοήματος. Είναι παγκοσμιοποιημένη η έρευνα, παγκοσμιοποιημένη η επιστήμη και έτσι πρέπει με δίκτυα να δράσουμε με κέντρο την αριστεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ να δώσω τον λόγο στον πρόσωπο της Κομισιόν για μια σύντομη παρέμβαση ή κάποιος άλλος εξ ονόματος Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που συμμετέχω στην πρώτη αυτή συζήτηση για το κοινό στρατηγικό πλαίσιο για την πράσινη βίβλο που έβγαλε η Κομισιόν πριν από λίγους μήνες. Από ό,τι βλέπω σήμερα από τη συζήτηση όλα τα θέματα τα οποία σας απασχολούν είναι αυτά που απασχολούν και εμάς. Οπότε συμπίπτουν οι σκέψεις μας κάποια σημεία που θα ήθελα να αναφέρω. Το ένα αφορά τον κατακαιρματισμό ή τη συνοχή ενό συγκεκριμένου τομέα πολιτικής. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να επιτύχουμε με την παρουσίαση του νέου πλαισίου, α το πούμε έτσι, να το πούμε πλαίσιο, εμεί ελπίζουμε να μην ονομαστεί πρόγραμμα πλαίσιο 8, αλλά να περιλαμβάνει και καινοτομία και βεβαίως και την πτυχή της εκπαίδευσης. Όταν λοιπόν εισαχθεί αυτή η νέα πολιτική, ελπίζουμε να είναι απλή. Αυτό είναι, αυτός είναι ο πρώτος μας στόχος. Δηλαδή να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα λειτουργεί για τον απλό ερευνητή που θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τους πόρους που προσφέρουμε και θα μπορεί με μια ματιά να αντιληφθεί ποιοι είναι οι στόχοι και τι προσπαθούμε να επιτύχουμε. Οπότε ελπίζω μπορούμε να, να μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό. Αυτό όσον αφορά και τον κατακριματισμό και τις συνέργειες με τις πολιτικές των κρατών μελών. Γιατί βεβαίως πρέπει να ξανασκεφτούμε τις ε, πολιτικές μας. Είμαστε σε καιρό κρίσης. Κάθε ευρώ πρέπει να μετράει. Πρέπει να υπάρχει προστιθέμενη αξία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μην γίνονται δύο φορές τέτοια πράγματα. Ή τέλος πάντων να μην υπάρχει άχρηστη αλληλεπικάλυψη. Να δούμε δηλαδή το τι γίνεται καλύτερα σε τοπικό και τι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όσον αφορά την υποεκπροσώπηση τώρα κάποιων περιφερειών της Ευρώπης. Αυτό αναφέρθηκε πολλές φορές. Χρειάζεται πράγματι εδώ πέρα συνεισφορά για να καταλήξουμε σε κάποιες ε, καλές λύσεις. Πρέπει να αυξηθεί η αριστεία σε κάποιες περιοχές και ξέρουμε ταυτόχρονα πως θα είναι δύσκολο για εμάς ε, να συμβιβαστούμε όσον αφορά το κριτήριο της αριστείας. Οπότε πρέπει να βρεθεί εδώ πέρα μια ισορροπία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γνωρίζουμε πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, οθούν την καινοτομία και πρέπει άρα να τις βοηθήσουμε. Ειδικά μέσα, ναι, ή ειδικά μέτρα. Αλλά δεν πρέπει να θεωρήσουμε πως ε, η απλοποίηση αφορά μόνο αυτές πρέπει να αφορά τους πάντες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να είναι εύκολη η πρόσβαση. Βεβαίως για τα ειδικά μέτρα να το δούμε αυτό, αλλά μην ξεχνάτε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σκέφτονται τοπικά. Πρέπει να μπορούμε να προσφέρουμε υπηρεσίες σε τοπικό επίπεδο. Και αυτό σημαίνει βεβαίως συνεργασία με το εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Τέλος, για το θέμα της απλοποίησης, η απλοποίηση είναι ένα στοιχείο κλειδί για την συζήτησή μας για το πρόγραμμα πλαίσιο 7. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε στο πρόγραμμα πλαίσιο 8. Έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε κάποιους κανόνες, ε, να πάμε σε ένα σύστημα που θα βασίζεται περισσότερο στην εμπιστοσύνη και αν χάσουμε αυτή την ευκαιρία θα είναι κρίμα για την έρευνα στην Ευρώπη. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Ματίας, ευχαριστώ. Ξέρω ότι έφτασε η ώρα της ψηφοφορίας, Πρόεδρε, αλλά σε κάθε περίπτωση θα ήθελα εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για όλες τις παρατηρήσεις και τα σχόλια που έκαναν. Χαίρομαι που έγιναν κάποια ζητήματα. και διαπιστώνω με τα χαράς ότι υπάρχει αρκετά ευρεία συνένεση σε σχέση με τα βασικά θέματα προσυζήτηση. Τώρα, ε, προφανέστατα θα υπάρξουν διχογνωμίες σχετικά με τον δρόμο που θα ακολουθήσουμε, αλλά ε, υπάρχει μια ευρεία συνενετική βάση, τουλάχιστον ως προς τον προσδιορισμό των βασικών προβλημάτων. Πολλοί συνάδελφοι σχολίασαν αυτό το δίπτυχο ε, ε, αριστεία συνοχή. Η αριστεία ναι είναι ένα κριτήριο αλλά όχι το μοναδικό και θα πρέπει ε, να συνδυαστεί με μια πολιτική που κατοχυρώνει ισότιμη πρόσβαση για όλους στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, όπως σας έλεγα και στην αρχική μου παρουσίαση. Οπότε, οι τέσσερις αυτές βασικές διαστάσεις της πράσινης βίβλου σε σχέση με το τι έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα, η απλούστευση της διαδικασίας, η χρηματοδότηση, τέλος πάντων για να μην επαναλαμβάνουμε αυτές οι τέσσερις βασικές διαστάσεις του στρατηγικού πλαισίου, μας βρίσκουν σύμφωνους αλλά θα πρέπει μετά από τη συζήτηση και θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους να προσδιορίσουμε σαφέστερα το πρόγραμμα πλαίσιο και τους επιμέρους τομείς τους, να προσδιορίσουμε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, ε, το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας και επίσης να οριοθετήσουμε επακριβέστερα το ρόλο των διαρθρωτικών ταμείων ως προς την έρευνα. Θεωρώ ότι η διασύνδεση αυτών των δύο ζητημάτων είναι ένα στοιχείο κλειδί για να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο, υπάρχουν, κυρίως ως προς τα κοινά ερευνητικά προγράμματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε τη σημασία της κοινής συμμετοχής δηλαδή των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα, κυρίως μιλώντας για επιστήμονες και επιστημονικά ιδρύματα που προέρχονται από ε, περιφέρειες ε, συνοχής. Ε, δεν θέλω να μακρηγορήσω, ήθελα μόνο να τονίσω ότι ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι το ΣΥΠ, το πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και κοινοτομίας. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να εκκρεμεί αυτό το ζήτημα. Οφείλουμε να δώσουμε μία απάντηση. Το αν θα ενσωματωθεί στο μελλοντικό πρόγραμμα πλαίσιο ή όχι θα το δούμε. Εγώ είμαι μάλλον κατά, αλλά προτίθεμαι να το συζητήσω μαζί σας κατόπιν διεθνή συνεργασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζεται διευκρίνηση και όριοθέτηση αυτών των δύο τομέων κυρίως ω προ τη σημασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Α, και κάτι που δεν αναφέρθηκε και θα ήθελα να το τονίσω, μία από τις μεγαλύτερε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ είναι η σχεδόν παντελής έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού εξειδικευμένου. Πρέπει να δώσουμε και σε αυτό ε, μία απάντηση. Για την απλούστευση και τα λοιπά δεν επαναλαμβάνω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι γιατί συμφωνώ. Ε, Εν κατακλείδη θα ήθελα να κάνω μία ε, τελευταία παρατήρηση. Χρειαζόμαστε την ε, ε, σωστή ισορροπία ανάμεσα στα μέσα που διαθέτουμε και τους στόχους μας, έναν από τους στόχους μας, δηλαδή πώς ακριβώς να αντιμετωπίσουμε και τις κοινωνικές προκλήσεις, πέρα από τις προκλήσεις στον τομέα της έρευνας. Και, επειδή ζούμε αυτή την οικονομική κρίση, δεν μπορούμε να δίνουμε μόνο τεχνολογικές απαντήσεις, χρειάζονται και κοινωνικές απαντήσεις και άρα χρειάζεται ισότιμη πρόσβαση όλων στα διαθέσιμα μέσα ε, Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα ε, κοινοτικά μέσα, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα εθνικά μέσα στη συνεργασία με άλλα κράτη-μέλη, αξιοποιώντας τις ε, ε, υποδομές που ήδη υπάρχουν, όπως είπε η συνάδελφος Κολάσκα Μπουμπίνσκα. Θα πρέπει λοιπόν η αριστεία να συνδυαστεί με την συνοχή, γιατί είναι άρετα συμφασμένες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σίγουρα θα επανέλθουμε πολλές φορές το ζήτημα σε μελλοντικέ ε, συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Τελειώνει το σημείο αυτό της ημερησίας διάταξης. Περνάμε στις ψηφοφορίες. Υποθέτω, συνάδελφοι, πώς έχετε φέρει όλοι τις κάρτες σας ε, για την ψηφοφορία. Να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Ποιος θεωρεί πως πρέπει να αυξηθεί ο φόρος στον ντίζελ. Ποιος θεωρεί... Όχι, όχι. Ας μην το πω και αυτό για τον κύριο Μπουτικόφερ καλύτερα. Λοιπόν, μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Λοιπόν, ποιο θεωρεί ότι πρέπει να ψηφίσουμε αρχή ψηφοφορία. Ε, μόνο να, να δουλέψετε με. Λοιπόν, πέρασε. Ωραία. Όλα εντάξει. Ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, υπάρχει μια πρόταση για μια αλλαγή στη σειρά εδώ πέρα. Ο συνάδελφος Κάλβιν ζήτησε να αλλάξει η σειρά των ψηφοφοριών. Αυτό γίνεται μόνο εάν το δεχτείτε. Θα ήθελε το σημείο 12 να ε, ψηφιστεί τελευταίο. Να το ξέρετε δηλαδή, αυτά δεν τα κάνει η γραμματεία, συνήθως οι συνάδελφοι. Δεν υπάρχουν αντίρρησεις, άρα έτσι γίνεται. Το 12 το ψηφίσουμε τελευταίο. Χάρη να με σημείο 8, ραδιοφωνικό φάσμα. Έχετε τον κατάλογο της ε, ψηφοφορίας. Ε, πρέπει να τα κάνουμε γρήγορα λοιπόν. Έχουμε πάρα πολλά. Προσέξτε λοιπόν. Έχουμε πολλές συμβαστικές τροπολογίες ευτυχώς. Συμβαστική ένα ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 unblock με την 3. 2 και 3 μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε στην 26 υπέρ. Κατά. Να το επαναλάβουμε. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 27 υπέρ. Ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι είναι. 27 υπέρ. Κατά. Ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία. 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 28 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Λοιπόν, συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 232 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 της ε, πολιτισμού υπέρ να επαληθεύσουμε την 233 άρχη της ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 28 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 234 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 236 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 23 αν ταυτόσημη. 31 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 239 υπέρ κατά αποχές δεκτή 240 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 του πολιτισμού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 241 υπέρ κατά αποχές δεκτή 243 υπέρ κατά αποχές δεκτή 244 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 245 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 246 υπέρ κατά αποχές δεκτή 248 και ΙΜΚΟ 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή ΙΜΚΟ 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 όχι 256 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή 265 υπέρ κατά αποχές δεκτή 266 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή Μήμικο 28 υπέρ. Κατά. Εποχές δεκτή. 271 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Κουλτ 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 πολιτισμό υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. όχι υπαριθμών 273 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 277 υπέρ κατά αποχές δεκτή 278 υπέρ κατά αποχές δεκτή 279 υπέρ κατά αποχές δεκτή 281 υπέρ κατά αποχές δεκτή 282 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται καταπίπτει συμβαστική εννέα να επαληθεύσουμε το δεύτερο μέρος. Ωραία. Τις... Το δεύτερο μέρος της ψηφοφορίας στις 2.82. Επαληθεύουμε λοιπόν. Ηλεκτρονικά. Κάποιος το ζήτησε. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. And... E Παραπάνω από το ΕΛΚ. Ωραία, πέρας. Απόρριπτοτε. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 298 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 300 υπέρ κατά αποχές δεκτή 304 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 44 υπέρ κατά αποχές κτή 346 υπέρ κατά αποχές δεκτή 349 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 351 υπέρ κατά αποχές δεκτή 357 υπέρ 357 υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή κουλτ 42 υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 358 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Κύριε Χεκμάρκ, για την 358 ε, υπήρχε και προφορική τροπολογία λοιπόν ε, δικτύων διανομής όπως ε, των υδάτων για να συμφωνεί με αυτό το οποίο πρότεινε η κυρία Τράουτμαν και η Λυπή. Δεν ξέρω αν συμπεριελήφθη. Ναι, βεβαίω, λέει ο πρόεδρο, είναι στο φάκελό σα. Το κάνω λίγο γρήγορα. Νόμιζα πω είναι σαφέ. Επειδή φοβήθηκα πω δεν ήταν αρκετά προφορική η τροπολογία, λέει ο κύριο Φεκμάρκ. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή. Κουλ 44 υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή. Ήμκο 39 υπέρ. Κατά Αποχέ. δεκτή. 367 υπέρ. Κατά Αποχέ. δεκτή. 368 υπέρ. Κατά Αποχέ. απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά Αποχέ. απορρίπτεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά Αποχέ. δεκτή. 381 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 383 υπέρ κατά αποχές δεκτή 382 υπέρ κατά αποχές ωραία ήμκο 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή 389 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 390 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 391 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 392 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 393 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 394 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 395 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 395 άρχη της ψηφοφορία and closed πέρας απορρίπτεται 396 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 398 υπέρ κατά αποχές 398 υπέρ κατά οι υπόλοιποι ποιο, ποιο λέμε 398 υπέρ μάλιστα κατά αποχές εγκρίνεται 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 399 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 400 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 51 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 52 υπέρ κατά Εποχέ. δεκτή 53 υπέρ κατά να το ξαναδούμε παρακαλώ 53 υπέρ κατά απορρίπτεται Ήμκο 1 υπέρ κατά εποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κουλτ 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ΙΜΚΟ 3 υπέρ κατά αποχές α, δεκτή 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή ΙΜΚΟ 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ 63 μας σχόλια υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται κουλ 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ήμκο 7 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ. Το ίδιο. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 75 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 76 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 90 υπέρ ε, 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 91 υπέρ πάω πολύ γρήγορα α συγγνώμη 20 20 σας τσεκάζει λοιπόν συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 91 υπέρ κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 97 υπέρ. Ναι. Τι. Κατά. Να επαληθεύσουμε. 97. Άρχιζε η σοφορία. Πέρασε. απορρίπτεται 6 υπέρ κατά δεκτή 98 υπέρ κατά εποχές δεκτή 99 υπέρ κατά εποχές δεκτή 7 υπέρ κατά εποχές δεκτή συμβαστική 22 υπέρ κατά α Λοιπόν, παριθμόν 9. 9. Υπέρ. Κατά που έχει 22 υπέρ. Κατά που έχει 117 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 118 υπέρ. καταπίπτει. Μάλιστα. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές 123 υπέρ. Κατά. Αποχές 11 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 125 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή κουλτ 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 135 υπέρ κατά 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή 135 υπέρ κατά αποχές δεκτή 134 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται κουλτ 14 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 136 υπέρ κατά εποχές δεκτή κουλτ 15 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 137 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 139 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κουλτ 17. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ψηφίζουμε τώρα. Συνολικά, ποιο είναι υπέρ. Ναι, ναι, ηλεκτρονικά καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται νομοθετικό ψήφισμα Ξανά πρέπει να ψηφίσουμε και το νομοθετικό ψήφισμα. Και άρχεται η ψηφοφορία. Κάποιοι λείπουν. Πέρας. Το, σχεδόν το ίδιο αποτέλεσμα. Συγχαρητήρια. Περνάμε από σημείο 9. Μέρκης τώρα, η κυρία Μέρκης. Συμβαστική 1 υπέρ. Πολύ γρήγορα πάω. Εντάξει, διάλειμμα. Yeah. Λοιπόν, συμβαστική 1 υπέρ. Κατά, αποχές, δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ κατά εποχές δεκτή συμβαστική 2 υπέρ κατά εποχές δεκτή Πενήντα έξι υπέρ κατά εποχές δεκτή 57 υπέρ κατά εποχές δεκτή λίγο ησυχία παρακαλώ 58 υπέρ. Κατά. Ναι, να υπαλληθεύσουμε. 58. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 67 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Να επαληθεύσουμε. 67. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. και εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 74 υπέρ. 74 ναι. Υπέρ. Κατά. Ναι. Τι τε κουραστήκατε. Λοιπόν. 74 υπέρ ξανά. Κατά. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Σαφές. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 103 υπέρ κατά αποχές δεκτή 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 111 υπέρ κατά αποχές δεκτή 112 χωριστή ψηφοφορία μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή 114 υπέρ να επαληθεύσουμε την 112 δεύτερο μέρος πέρας ένας παραπάνω από το ΕΛΚ εντάξει δεκτή 114 υπέρ Κατά. Αποχές δεκτή. 116 πέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 129 υπέρ. Κατά αποχές 130 υπέρ κατά αποχές συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 11 α υπέρ κατά αποχές δεκτή 137 υπέρ κατά αποχές δεκτή 138 υπέρ κατά αποχές να επαληθέψουμε 138 άρχεται ψηφοφορία και πέρας και εγκρίνεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 151 υπέρ κατά αποχές δεκτή 152 υπέρ κατά έχει δεκτή 153 υπέρ κατά έχει δεκτή 154 υπέρ κατά έχει δεκτή 155 υπέρ κατά έχει δεκτή 157 υπέρ κατά 157 επαναλαμβάνουμε υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 159 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 161 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 165 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 166 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 167 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 177 υπέρ κατά αποχές δεκτή 178 υπέρ κατά αποχές δεκτή 179 υπέρ κατά αποχές δεκτή 180 υπέρ κατά αποχές δεκτή 181 υπέρ κατά αποχές δεκτή 184 υπέρ κατά αποχές δεκτή 186 υπέρ κατά αποχές δεκτή 187 υπέρ κατά αποχές δεκτή ναι να επαληθεύσουμε 187 υπέρ και πέρας και δεκτή συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 191 υπέρ κατά αποχές δεκτή 193 υπέρ κατά αποχές δεκτή 195 υπέρ κατά αποχές δεκτή 196 υπέρ κατά αποχές δεκτή 197 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. 197. Άρχιτε η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική 20. Υπέρ. Κατά. Εποχές δεκτή. 201 υπέρ κατά αποχές δεκτή 202 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 209 υπέρ κατά αποχές δεκτή 213 υπέρ κατά Εποχές. Απορρίπτεται. 214 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. 214. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τεκτή. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Τεκτή. 222 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 226 υπέρ. Κατά. 226 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. 227 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 229 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεκτή. 230 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεκτή. 231 υπέρ. Κατά. Να το ξαναδούμε. 231 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 232 υπέρ. Κατά. Δέκτη. Συμβαστική 26 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 238 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 239 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 27 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 28 α υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 29 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 252 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 30 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 259 υπέρ κατά αποχές δεκτή 260 υπέρ κατά ξανά 260 υπέρ κατά να επαληθεύσουν την 260 άρχεται η ψηφοφορία και πέρασε απορρίπτεται συμβιβαστική 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 270 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 271 υπέρ κατά αποχές δεκτή 272 υπέρ κατά αποχές δεκτή 273 υπέρ κατά αποχές δεκτή 274 υπέρ κατά αποχές δεκτή 32 συμβαστική υπέρ κατά αποχές δεκτή 290 υπέρ κατά αποχές δεκτή 291 Ναι, να επαληθεύσουμε τη 290 άρχη τη ψηφοφορία πέρας και δεκτή 291 υπέρ κατά αποχές δεκτή 292 υπέρ κατά αποχές δεκτή 293 υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 297 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 298 υπέρ κατά αποχές δεκτή 299 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να επαληθεύσουμε 299 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Ναι, δεκτή, σαφώς. 300 υπέρ. Κατά. Δεν ξέρω. Λοιπόν, 300 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 301 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβασική 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 υπέρ κατά 36 υπέρ. Κανείς. Ξέχασα κάποια. Α, με συγχωρείτε. Συμβιβαστική 35, η πιο σημαντική από όλε. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Οπότε, πού πάμε τώρα. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τριάντα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. αποχέ δεκτή. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 40 υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή. 41 υπέρ. Κατά. Αποχέ. απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή. 2 υπέρ. Κατά. Αποχέ δεκτή. Δεν μπορούμε να τις κάνουμε όλες μαζί. 3 έως 7. 3 έως 7 μαζί. Ωραία. Υπέρ. Κατά. Ωραία. Δεκτές. Τώρα, ένα ίντα υπέρ. Unblock. 1 έως 6 ποιος είναι υπέρ. Όχι. Γίνεται ή όχι από την 1 έως την 6 τη ΣΥΝΤΑ. 1 έως 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Οπότε είναι τα 10 υπέρ. Α, 8, 8, με συγχωρείτε. Υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 10 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 12 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 14 έως 16 πάνε μαζί, όχι. 14 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Α, γινότανε. Ε, Τη Επιτροπή Αποσχόληση. Μπορούμε μετά το 2 έως 5 να τις κάνουμε μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Λοιπόν, και άλλες μαζί. 7, 11, 12, 14, 15, 17. Μπορούν να γίνουν μαζί. Ωραία, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εποχές δεκτές. 19 δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 20 με 23 μπορούμε. Μαζί υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές. 26 υπέρ κατά αποχές δεκτές 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή να υπαλληθεύσουμε ωραία 27 άρχεται η ψηφοφορία ένας παραπάνω από το ΕΛΚ πέρας και δεκτή του περιβάλλοντος τώρα 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 να πάνε μαζί. Μέχρι την 9. Μέχρι την 7. 1, 4 και 7. Ποιος είναι υπέρ. Όχι. 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 8 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 8 υπέρ 9 με συγχωρείτε 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 με 22 μπορούμε να τα κάνουμε μαζί 19 έως 22 μπλοκ. Ναι. Υπέρ. Τι, τι τρέχει τώρα. Καλύπτονται. Α, λάθος κατάλογο έχω. 20 και 21. 20 και 21 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ε, είναι ο βραδινό κατάλογο χαό και αλλάζει με την ώρα 25. Πρώτο μέρο υπέρ. Κατά Αποχέ, απορρίπτεται. 26 υπέρ. Α, συγγνώμη, πάλι λάθος κατάλογος. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. Να επαληθεύσουμε 27. Α, έρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Και εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. 29 υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και έγκρινεται. 30. 30, 31 και 32 να τις κάνουμε μαζί. Όχι. 30 υπέρ. Κατά. Εποχές. Δεκτή. 31 υπέρ. Κατά. Εποχές. Δεκτή. 32 υπέρ κατά νομίζω γίνεται δεκτή καμία αντίρρηση, ωραία ε, κύριε εντάξει μου επιτρέπει ο κύριος Μπιτικόφερ εντάξει επόμενη τρία Ίμκο από 7 έως 11 όχι 7 έως 9 Ούτε αυτό. 7 έως 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτές. 10 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 11 υπέρ. Κατά Αποχέ δεκτή. 17 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 18 πρώτο μέρος. Είναι, εγώ έχω το χθεσινό βραδινή λίστα. Λοιπόν, τρία τη Ρέγκη. Ναι. Είπα αριθμό τρία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Δεκτή. Τέσσερα. Τέσσερα, πέντε, έξι μαζί. Τέσσερα, πέντε, έξι μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. δεκτές. Οχτώ και εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. δεκτές. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 και 18 μαζί υπέρ όχι 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 και 22 υπέρ κατά αποχές δεκτές Κουλτ 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 7 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 8 υπέρ. 9 και 11 όχι 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά Να επαληθεύσουμε. 17 άρχιδη ψηφοφορία. Πέρας. Και... απορρίπτεται. 18 υπέρ. 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. ABC να τις ψηφίσουμε μαζί. Όχι. Α υπέρ κατά αποχές δεκτή. Β υπέρ κατά αποχές δεκτή. Γ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δ υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δύο υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τέσσερα υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά ξανά με ηλεκτρονική ψηφοφορία την 5 άρχη της ψηφοφορία ε, closed. πέρασε και δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά ξανά 7 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 7 άρχεται η ψηφοφορία και πέρασε και δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ωραία 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή ορίστε τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική άρχεται πέρας ένα παραπάνω από το ΕΛΚ. Και... Ωραία, συγχαρητήρια. And Ευχαριστώ τους συναδέλφους που έκαναν τις συμβαστικές τροπολογίες. Περνάμε στο σημείο 10. Ακόμα έχουμε. Κύριε Οντή. Two amendment the green time. Oh mein Gott, multitasking. Amendment 3, Zustimmung. 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 6 υπέρ, κατά, αποχές. Και πάλι, 6 υπέρ, κατά. Απορρίπτεται 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 19 Επίσης προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 36 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ε, συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 ε, συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται. Η 17 συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 77 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Budget. 3. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά Αποχέ δεκτή 56 υπέρ κατά Αποχέ δεκτή 72 υπέρ κατά Αποχέ δεκτή 72 αν δεν επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία Closed. Mr. Κύριε Μπουτικόφερ, Ψηφίστε. Καμία αντίρρηση σήμερα δεν έχετε. Μάλιστα. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Και τι γίνεται τώρα. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 83 υπέρ Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. 83. 83 είπαμε. Και... Απορρίπτεται. 88 υπέρ. Ευχαριστώ. Κατά. Ναι. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 96 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 97 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 99 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ. Συμβιβαστική 10. Ματίας. <coughs> Λάθος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πριν να ψηφίσουμε αυτή τη συμβαστική θα ήθελα μόνο να σας πω ότι παρότι μέσα στην, στον κατάλογο φαίνεται αυτή η τροπολογία που κατέθεσα εγώ και σβήνει το μικρόφωνο της ομιλήτριας, δεν ακούσαμε τη συνέχεια. Ζητώ συγγνώμη, μου σβήσε το μικρόφωνο. Λοιπόν, πριν ψηφίσουμε αυτή την, ε, την συμβαστική τροπολογία και παρότι στον κατάλογο ε, φαίνεται ότι η τροπολογία 114, η δικιά μου δηλαδή, ότι καλύπτεται από τη συμβαστική, μετά από συμφωνία με τον εισηγητή τον κύριο Οντή, αποφασίσαμε ότι πρέπει χωριστά να ψηφίσουμε την τροπολογία μου, διότι δεν καλύπτεται από αυτή τη συμβαστική σχετίζεται η τροπολογία με, ε, με, την, ε, με τον επισφαλή χαρακτήρα, αν θέλετε, των ε, θέσεων ερευνητών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλάμε για τη συμβαστική 10 αυτή τη στιγμή. Πάει, 9 ψηφίσαμε. Ακριβώς, ακριβώς, γιατί 10 είπαμε, ε, οι 110, 113, 114 και διάφορε άλλε καλύπτονται από αυτή τη συμβαστική τροπολογία. Όσως μιλάω για την 114 και μετά από σύμφωνη γνώμη του εισηγητή του κ. Ντί, αποφασίσαμε ότι θα ψηφιστεί χωριστά αυτή η τροπολογία συγκεκριμένα. 114 δεν καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία και σα λέω σχετίζεται με την επισφαλή χαρακτήρα των ε, ερευνητικών θέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κύριε Ντί, συμφωνείτε λέμε ότι λυπούμεθα που είναι επισφαλής ο χαρακτήρας αυτών των θέσεων ερευνητών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι πολύ καλή η διατύπωση, πολύ κομψή, αλλά ε, για να επιτύχουμε το συμβασμό, ναι, συμφωνώ. Συν Ωραία. Συμβαστική 10 χωρίς το 114 ποιος είναι υπέρ. Ευχαριστώ, κατά, εποχές δεκτή. 114 χωριστά, υπέρ κατά αποχές δεκτό 116 υπέρ κατά αποχές δεκτό 118 υπέρ κατά αποχές δεκτό 119 υπέρ κατά αποχές δεκτό συμβαστική 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 143 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 148 υπέρ κατά αποχές δεκτό. 150 υπέρ 150 υπέρ. Εκατόν πενήντα. Αυτοί είναι όλοι. Κατά. Ε, αν θέλετε, θα επαληθεύσουμε. Άρχιε τη ψηφοφορία. Για το 150. Yeah, yeah. And check closed. Πέρας. Closed. And, and adopted. Δεκτή. Καταπίπτει, καταπίπτει. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 164 υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. 166 υπέρ. Κατά. 166 υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. 167 υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. 168 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 170 υπέρ κατά αποχέ δεκτή συμβαστική 15 υπέρ κατά απόχέ δεκτή συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχέ δεκτή 209 υπέρ κατά δεν μπορώ να καταλάβω 209 υπέρ κατά αποχές δεκτή 213 υπέρ κατά αποχές δεκτή 214 υπέρ κατά αποχές δεκτή 215 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 216 υπέρ κατά αποχές δεκτή 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 217 να επαληθεύσουμε παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Δεκτή. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 238 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε 238 άρχεται η ψηφοφορία πέρας δεκτή 239 υπέρ κατά αποχές δεκτή 240 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 278 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 283 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 285 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Budget όχι. 286 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 287 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 290 υπέρ Κατά. 2,90 υπέρ. Κατά. Δεκτή. 291 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 292 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 293 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 297 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 298 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 302 υπέρ κατά αποχές δεκτή 303 υπέρ κατά αποχές δεκτή και τελική ψηφοφορία Α, κύριε Οντή, με συγχωρείτε. Πρόεδρε, αν δεν κάνω λάθος, αλλά θα ήθελα να το εξακριβώσει η γραμματεία μου, φαίνεται ότι δεν ψηφίσαμε την συμβαστική 17. Δεν είναι στον κατάλογο της ψηφοφορίας. Κάνω λάθος, μου λέτε. Θα μπορούσατε να το εξακριβώσετε. Μου φαίνεται ότι δεν ψηφίσαμε τελικά τη συμβαστική 17. Πρόκειται για την ισότητα των ευκαιριών των δύο φίλων. Είναι αρκετά σημαντική. Μπορείτε να το εξακριβώσετε. Εγώ νομίζω ότι το έχουμε ψηφίσει όλοι. Ναι. Zugestimmt. Zugestimmt. So, damit können wir jetzt ganz ruhig in die Abstimmung gehen. Final vote. Ωραία, μπορούμε να πάμε στην τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Και πέρασε. Συγχαρητήρια. Περνάμε άρα στην έκθεση ΡΕΜΕΚ στην επόμενη. Ε, μα, ε, αυτοί αλλάζουν συνεχώς και εγώ συνεχίζω ίδιος. Είναι αδικαία, λέει ο πρόεδρος. Οπότε τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 υπέρ κατά να το ξαναδούμε. Υπαριθμόν 3 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε την 3. Άρχεται η ψηφοφορία. 3. Πέρας. Εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 4 α υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ ε, μέρος πρώτο με συγχωρείτε υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτό 19 υπέρ κατά αποχές δεκτό 23 υπέρ κατά αποχές δεκτό 24 όχι 25 υπέρ κατά αποχές απορρίφτεται 26 υπέρ κατά αποχές δεκτό 30 υπέρ κατά αποχές δεκτό 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτό 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 υπέρ κατά αποχές δεκτό 41 υπέρ κατά αποχές δεκτό 44 υπέρ κατά αποχές δεκτή 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή και περνάμε 48-49 μπλοκ υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές δεκτή 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική άρχεται πέρας Πέρασε. Δεκτή. Συγχαρητήρια. Περνάμε στο σημείο 13. Ρόντι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή, συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή, Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ υπέρ κατά 3 επαλήθευση να επαληθεύσουμε Can I close? No. Πέρας. Δεκτή. Γίνεται δεκτή η τρία. Εντεκά Τώρα, σωστά. Δώδεκα. Δώδεκα. Η τρία έγινε δεκτή. Και περνάμε στην τροπολογία 12. Τροπολογία 12. Ακριβώς από κάτω. 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 14 υπέρ. Κατά αποχές Πώς Επόμενη, 17. Okay. Ε, ε, Όταν αρχίσαμε, δεν το υπενθυμίσατε. Τέλος πάντων, επικράτησε σύγχυση μετά και θα ήθελα να προτείνω να ξαναρχίσουμε την ε, ψηφοφορία. Sorry. Yeah, yeah, yeah. Von von vorne? Von ganz vorne, von heute Morgen? According to... Από πού να ξαναρχίσουμε. Μα, ε, συγγνώμη, βάσει της σειράς που έχει προβλεφθεί, το ίδιο χαρτί έχουμε, αλλάξαμε. Κανείς δεν υπενθύμησε ότι άλλαξε αυτή η σειρά και γι' αυτό δημιουργήθηκε η σύγχυση. Hm, ακολουθήσαμε τον κατάλογο. <laughs> Τι, από την αρχή θα ξαναπάρουμε τώρα να ξαναψηφίσουμε όλη την έκθεση. Συγγνώμη, τη συμβαστική τρία, αυτή συζητούσαμε τώρα. Λοιπόν, ξανά, συμβαστική τρία. 3. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συμβαστική 3. Ψηφίστε παρακαλώ. Για την έκθεση ρόντε. Τώρα, αυτό, ούτε αυτό δεν έχουμε ξεκαθαρίσει. Now we are... Hey, ladies and gentlemen, can we fasten your seatbelts? Can we... Προσδεθείτε, κυρίες και κύριοι, θα απογειωθούμε. Λοιπόν, έκθεση Ρόντε. Συμβαστική 3. Βλέπετε τι γράφει ο κατάλογος. So, jetzt machen wir noch mal, jetzt aber bitte, ladies and gentlemen. Σας παρακαλώ. Συμβαστική τρία της έκθεσης ρόνται με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Τελευταία φορά θα το πω. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Τα ίδια. Δώδεκα. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Σημαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ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 απόχες εγκρίνεται 71 υπέρ ε, ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία πέρας 71 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 72 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία, με ηλεκτρονική ψηφοφορία βεβαίως. Enclosed. Πέρας. And adopted. Εγκρίθηκε, είναι σαφής η πλειοψηφία. Συγχαρητήρια. Ja, muss ich das wissen? Ja, weil die um Bleiben Sie, bleiben Abstimmung hier. So. 14. New Trade Policy for Europe. πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση Στρατηγική 2020. Er Δεν μπορώ να το προφέρω το όνομά του. Ε, Βοηθήστε με. What's the Πώς ακριβώς το προφέρετε το όνομά σας, αλήθεια. Τρόμος. Mm. Άμα εξασκηθείτε θα τα καταφέρετε καλύτερα. Ε, προφέρετε, πολύ ωραία. Η έκθεση του κυρίου Γκζιμπ λοιπόν. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 31 σε δύο τμήματα, το πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται, το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει το δεύτερο τμήμα, Πρόεδρε. Ζητά συγγνώμη ο Πρόεδρος. Ε, καταπίπτει το δεύτερο τμήμα γιατί εγκρίθηκε συμβαστική 2. Τώρα η 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ε, ε κατά τμήματα 17 πρώτο υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται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 κατά αποχές εγκρίνεται ε, κατά τμήματα η 30 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 υπέρ κατά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 Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Με μία μόνο αποχή και δύο ψήφους κατά εγκρίθηκε. Nein. Jetzt kommt Nummer 12. Kollege Vidal Quadras. Ο συνάδελφος Βιντάλ Κουάντρα. Ένα διαδικαστικό έχω κύριε Πρόεδρε. Ρωτήσατε πώς προφέρετε το επώνυμο του κυρίου Γκζιμπ. <laughs> Μα ένα επώνυμο με πέντε σύμφωνα χωρίς εντά <laughs> είναι για μας τους μεσογειακούς δυσμενής διάκριση. Εις βάρος μας οπότε θα πρέπει τώρα να κάνουμε μια αναθεώρηση της συνθήκης. Θέλουμε αντιστάθμιση, αποζημίωση. Δεν έχουμε χρόνο, τώρα μην βαθύνουμε το σημείο, έτσι. Ε, κοιτάξτε, θα εμβαθύνω λίγο. Ε, ο Φιλανδός συνάδελφος ε, θα ήθελε επίσης αντιστάθμιση. Κοιτάξτε, ε, σε διάφορες γλώσσες ε, υπάρχουν πολλά τέτοια σύμφωνα. Άμα θέλετε να το συζητήσουμε κατηδίαν σήμερα το απόγευμα, Πρόεδρε. Δεν είναι εδώ συνάδελφος Κάλφιν. Good, trotzdem, es geht los. Punkt... Ξεκινάμε. Ε, τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 44 και 9 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 45 και 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Α, κατέπεσε. 48 τότε υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται 50 υπέρ. Συγγνώμη. Έχει καταπέσει 50 λέει ο πρόεδρος. 51 υπέρ. Κατά τμήματα ψηφοφορία σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Ηλεκτρονικός έλεγχος Α, το δεύτερο τμήμα κάνουμε. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 51, το δεύτερο τμήμα, παρακαλώ. And closed? Πέρας. Oh, rejected. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγγνώμη, υπέρ, ξανά, κατά αποχές εγκρίνεται, 75 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 76 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 77 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 78 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 79. Ε, συγγνώμη, έχει καταπέσει υπέρ, κατά απόχέ. απορρίπτεται, 80 80 και 82 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται 83 υπέρ. Την 80 θέλετε, έλεγχο. Ωραία. Ωραία, 80 82 ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ. And check, yeah, closed. Πέρας. Σχεδόν το κατάφερες, σε 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 20 και 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται 21 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία ηλεκτρονική άρχεται παρακαλώ ψηφίστε ψηφίστε παρακαλώ and closed πέρας mm. and adopted εγκρίθηκε και τώρα. Συγχαρητήρια, ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για τη φοβερή σας πειθαρχία. Μια χαρά τα πήγαμε, μια μισή ώρα μόνο ψηφίζαμε. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ για τη βοήθειά σας και τώρα, εάν αποχωρήσετε όλοι όσοι έχουν δουλειά να κάνουν έτσι μόνο, αν αποχωρήσετε λοιπόν γρήγορα μπορούμε να συνεχίσουμε κι εμείς. Το επόμενο σημείο είναι η συνολική προσέγγιση όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Giles, Chichester, παρακαλώ λίγη ησυχία. Μόνο ο κύριος Τσίτσαστερ θα μιλάει τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τώρα, εάν επιμένει κανείς να μείνει ή αν μιλάει, θα τους κανονίσω εγώ προσωπικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται εγώ για κάποια έκθεση που αφορά το θέμα της προστασίας των δεδομένων και έχουμε συντάξει μια ευσύνοπτη έκθεση, γνωμοδότηση που παρακαλώ συνάδελφοι να την εγκρίνετε. Θα ήθελα να σας τονίσω τι θέλουμε να πούμε. Στην ουσία θέλουμε να μην έχουμε γραφειοκρατία, μην βαρύνουμε υπερβολικά τις επιχειρήσεις με τυπικότητες και πιο συγκεκριμένα προστατεύσουμε τις ΜΜΕ από αυτό ε, και να μην βαρθούν επομένω με την νομοθεσία μας. Ε, ελπίζω δε, συνάδελφοι, ότι θα συμφωνείτε. Θέλουμε η Κομισιόν να προσέξει τις παραγράφους 1, 2 και 3. Διότι έχουν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία όσον αφορά ακριβώς την επίτευξη του στόχου μας. Η παράγραφος 5 αφορά το θέμα της προστασίας του ιδιωτικού βίου. Τώρα, λέει η Κομισιόν Privacy by Design ε, ιδιωτικό βίο προστασία του βίου μέσω σχεδίου. Μα τι εννοεί ακριβώς, γιατί εδώ πέρα επιδέχεται πολλές ερμηνείες αυτό ο όρο αυτή η φράση. Τώρα, στο 6, παράγραφος δηλαδή 6, Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μελετήσει τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων περισσότερο αυτό παρά την υποχρέωση λογοδοσίας όπως έχει αναφέρει και στο 7 επανερχόμεθα στο θέμα του να μην έχουμε υπερβολικές τυπικότητες που να επιβαρύνουν τις ε, επιχειρήσεις και τους εμπλεκόμενους. Αυτά πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά να ακούσω τις απόψεις των συναδέλφων και εδώ βάζω τελεία. Well, or shall I carry ή όχι. Να συνεχίσω μέχρι να σταματήσει την κουβεντούλα ο κύριος Λάγκεν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο πρόεδρος. Ευχαριστούμε εμείς κύριε Τίλιστερ. Και τώρα ε, ο κύριος Χρόντο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Τίτσεστερ. Για όσο μας εξηγήσατε, για όσο έχετε γράψει, το θέμα είναι περίπλοκο γιατί σε κάθε πρόοδο της τεχνολογίας θα πρέπει κανείς να εξασφαλίζει ότι υπάρχει αντίστοιχη προστασία των δεδομένων. Ε, να μην είμαστε πάντοτε πίσω όσον αφορά τις ε, πρόοδους τεχνολογίας, να μπορούμε επομένω να παρακολουθήσουμε και να μην χάνουμε το τρένο της τεχνολογίας. Η ψηφιακή ατζέντα ξέρουμε ότι προχωράει και θα πρέπει επομένω να διευκολύνουμε τις ΜΜΕ. Δεν θέλουμε σε κράτη-μέλη να υπάρχουν διαφορές ε, όσον αφορά αυτές τις ε, υποχρεώσεις τις διοικητικές. Πάντως εδώ δεν εμπλέκονται μόνο οι ΜΜΕ. Έχουμε και τα κοινωνικά δίκτυα τα οποία επίσης έχουν επιπτώσεις. Επομένως, να δούμε πώς οι χρήστες θα την χάνουν προστασίας του ιδιωτικού τους βίου και των ε, προσωπικών δεδομένων τους. Εκεί όπου χρειάζεται να δίνουν κάποιες πληροφορίες θα πρέπει επομένω να εκτενήσουμε την ε, διατύπωση στις σχετικές παραγράφους, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι κάποια νέα δεδομένα, όπως κάποια γενετικά δεδομένα τα οποία στο μέλλον θα χρησιμοποιούνται, θα καλύπτονται από αυτή τη ρύθμιση και να μην ε, προσπαθούμε εκ των υστέρων να προλάβουμε τις εξελίξεις. Επομένως, η εναρμόνιση εξοικονομεί χρήματα, δεν θα πρέπει η, αντίθετα να συνεπάγεται δαπάνες. Σύμφωνο βέβαια μετά όσο έχει πει ο συγητής, θα πρέπει να βρεθεί η κατάλληλη ε, ισορροπία της ρύθμισης στην Επιτροπή μας και έτσι να καλύπτονται όλοι και όχι μόνο η ΜΜΕ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Νίμπλερ, και εσείς ε, στην Επιτροπή σας έχετε αναλάβει να προωθήσετε το θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει κυρία Νίμπλερ. Όχι, όχι, πρόεδρε, δεν εκπροσωπώ την ε, Επιτροπή. Α, ναι, ναι, ναι, η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχει δίκιο, πρόεδρε, έχει δίκιο. Όχι, νόμιζα. Ήταν, έφταιγε η Επιτροπή Δημοκρατικών Ελευθερίων. Ε, με μεζάλισαν οι ψηφοφορίε. Ευχαριστούμε επομένω για την έκθεση και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σωστό το ότι εξετάζουμε εδώ ε, το αποτέλεσμα στη δράση των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το πρέπει να ζητηθεί κι άλλο. Τα ακούσαμε και χθε από την Ελικρού στην Επίτροπο που μα είπε ότι του ε, μέσου επόμενου μήνε πρόκειται και αυτή να μελετήσει το θέμα τη ψηφιακή τεχνολογία, τη ψηφιακή ατζέντα και μα είπε ε, ότι το cloud computing θα είναι μια στρατηγική που θα επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση αμέσω επόμενου μήνε. Άρα θα πρέπει και η δική μα επιτροπή να προσέξει το τι θα γίνει με την προστασία των δεδομένων. Πώ θα την εξασφαλίσουμε. Συμφωνώ βέβαια με όλου του προλαλήσαντε είναι το θέμα σημαντικό. Να το παρακολουθήσουμε. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την διεθνή διάσταση τη υπόθεση προστασία των δεδομένων. Να δούμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο όσον αφορά τα δεδομένα. Αν θέλουμε να έχουμε το ίδιο επίπεδο προστασία των δεδομένων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ρυθμίσουμε για το τι γίνεται με τα δεδομένα τα οποία ζητούνται εκτός Ένωσης. Και δεν είναι θέμα πίστης, εμπιστοσύνης, καλή ε, θέληση με τον συνομιλητή μας. Πρέπει θεσμικά να υπάρχουν οι έλεγχοι και η κατάλληλη δομή του πλαίσιου ασφάλειας, ας πούμε όπως συμφωνήθηκε με τις ΕΠΑ. Να δούμε επομένω όσοι έχουμε συμφωνήσει, εάν είναι εξυγχρονισμένα, ενημερωμένα, επικαιροποιημένα, γιατί χρειάζεται να υπάρχει τέτοια ρύθμιση προ των δεδομένων. Θα πρέπει να δούμε επίση τι καλύπτεται, ποια δεδομένα καλύπτεται από αυτή τη ρύθμιση κλπ. Κάθε φορά που έχουμε μεταφορά δεδομένων, να δούμε αν ο πολίτη προστατεύεται, τι συνέπειες υπάρχουν. Επίση τώρα, όσον αφορά αυτήν την προστασία ιδιωτικού βίου by design που λέμε, με, με σχέδιο. Τι εννοεί. Μέσω σχεδίου. Τι εννοεί. Έχει δίκιο ο Τσίτσεστερ. Τι, τι, τι πάει να πει αυτό. Άρα να κάτσουμε και να εξασφαλίσουμε το πώς. Η αυτόματη ρύθμιση ούτω υπήν θα είναι η προστασία του ιδιωτικού βίου, ο σεβασμό του ιδιωτικού βίου από τι εταιρείε. Τέλο πάντων, έχετε δίκιο. Χρειαζόμαστε περισσότερα στοιχεία. Τι θα πει αυτό. Ποιε είναι οι συνέπειε σε πανευρωπαϊκό, σε ενωσιακό επίπεδο, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τον κόσμο, με του νέου που χρησιμοποιούν κάθε μέρα την τεχνολογία. Να ξέρει ο κόσμο τι συμβαίνει, πού πάνε τα δεδομένα του. Αξίζει να γίνει επίση μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωση. Τα δέκα μέλη να μην κάνουν το καθένα ό,τι θέλει. Θέλουμε ενωσιακή προσέγγιση. Έτσι, να βελτιωθεί το επίπεδο της ενημέρωσης και επομένως θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και στο μέλλον. Θα σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Κομίνσκα, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρώτα-πρώτα, να ευχαριστώ τον κύριο Τσίτσεστερ για τη γνωμοδότηση. Το μήνυμα αυτό το οποίο έτσι στέλνουμε ως αφορά την δεδομένων είναι το σωστό. Έτσι θα πρέπει να υπάρχει ισόρροπη ρύθμιση και επομένω θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ προστασίας ιδιωτικών ε, ε, και προσωπικών δικαιωμάτων και από την άλλη μεριά εύρυθμη λειτουργία των ε, επιχειρήσεων χωρίς να τις βαραίνει η γραφειοκρατία και τα, τα, τυπικότητες. Να δούμε τι πρέπει να αλλάξουμε τι πρέπει να προσθέσουμε στο κείμενο. Νομίζω θα πρέπει να είμαστε πιο ανοιχτοί όσον αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας ε, διότι νομίζω ότι δεν γίνεται αυτό τώρα με αυτήν την οδηγία. Να επισημάνουμε στην Κομισιόν ότι θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική με τις καινούργιε αρχές. Να, να, να μόνο ότι πραγματικά χρειάζεται. Δοκιμές. Να γίνονται δοκιμές. Όπου χρειάζονται. Τώρα, όσον αφορά αυτά τα κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα, ποια, ποια είναι η έννοια της συνένεσης, ε, σε ποια ηλικία θα πρέπει να δίνεται, ε, τι γίνεται όσον αφορά την ε, κατοικία, διεύθυνση. Είναι, είναι δύσκολο το, το, να επισημανθούν αυτά. Τώρα κάτι άλλο, όσον αφορά την υποχρέωση λογοδοσία συμφώνω στον νόμο θα πρέπει να αναζητηθεί μια λύση σε σχέση με το ποιο είναι ο υπόλογο, ποιο είναι υπεύθυνο όταν έχουμε πολλαπλότητα συλλογή δεδομένων. Γιατί πάρα πολλέ φορέ έχουμε περισσότερου από έναν αποδέκτες δεδομένων. Τώρα επίσης ε, για αυτές τις ε, σφραγίδες, τα, τα, τα, πιστοποιητικά θα πρέπει εδώ πέρα να εξασφαλίσουμε ε, ότι υπάρχει σωστικός έλεγχος και δεν μπορεί ο καθένας να, να κάνει copy-paste αντιγράφει τέλο πάντων από τη μία ιστοσελίδα στην άλλη, ε, από το ένα παράθυρο του υπολογιστή στο άλλο, τα δεδομένα. Την ανταλλαγή δεδομένων να δούμε μεταξύ των ε, νομικών προσώπων και να υπάρχει σε όλη τη διαδρομή δυνατότητα ελέγχου. Επίσης να δούμε τι τροποποίηση στα δεδομένα ε, είναι εφικτή στη διαδρομή διαβίβαση των δεδομένων. Να μπορεί κάθε φορά να, να τρέξει κανένα στην πηγή των πληροφοριών. Επίσης ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να μας ξεκαθαρίσει ποια είναι η σχέση μεταξύ προστασίας δεδομένων και κάποιο είδους ε, δυνατότητας άσκησης ομαδικών αγωγών. Δεν είμαι κατά. Όμως θα πρέπει η Κομισιόν να ξεκαθαρίσει τη θέση της και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Εκ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον Giles Chichester για την έκθεσή του. Θεωρώ ότι κατάφερε να συγκεράσει τα επιμέρους ε, συμφέροντα εύστοχα. Δυστυχώ, έγινε κάτι δυσάρεστο. Επί πολύ χρόνο παραμιλήσαμε θέματα όπως προστασία ιδιωτικού βίου, ασφάλεια, ακαιρεότητα. Τα συναφή δικαιώματα επομένω. Το σωστό είναι να δούμε πώς θα βρεθεί μια κοινή πορεία που θα συγκεράζει, θα συγκεράζει και το στόχο μας με τις ε, λογικές δαπάνες, με τα ατομικά δικαιώματα. Η ασφάλεια είναι πάρα πολύ βασικό, αλλά ε, και οι δαπάνες επίσης θα πρέπει να συνυπολογιστούν. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όσες εύστοχες ρυθμίσεις περιέχει το κείμενο του Giles. Νομίζω ότι είναι εύστοχη επίσης η ρύθμιση αυτής της privacy by design προστασία ιδιωτικού βίου με το σχέδιο. Το ίδιο αφορά και η αποθήκευση δεδομένων των φυσικών προσώπων. <coughs> Τόσα καιρότητα πάντως υπάρχουν κίνδυνοι και είναι πάρα πολύ σημαντική από πλευρά αυτών που επιδέξει. χειρίζονται το διαδίκτυο. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι δαπάνε γίνονται από πλευρά φυσικονομικών προσώπων χωρίς να έχουμε ε, τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την ασφάλεια. μένουν. και εδώ τα λέει καλά ο Giles. Πάντως θα πρέπει να ζητηθεί και άλλο το θέμα προς την κατεύθυνση που σας εξήγησα. Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν υπάρχει εδώ εκπρόσωπος της Κομισιόν ή όχι. Τέλος πάντων. Τζάιλς, θες εσύ το λόγο. Τσίτσεστε. Α, όχι, μισό λεπτό. Α, και, ε, μόλις ήρθα και αν θέλετε μπορώ να σας μιλήσω αργότερα. Λευκό Επιτροπή. Ευχαριστούμε την Επιτροπή, σε ευχαριστώ και τον εισηγητή. Δεν έχω τίποτα συγκεκριμένο να σα πω γιατί όλα αυτά τα οποία αναφέρατε τα διεξερχόμεθα στην έκθεση επιπτώσεων και θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το θέμα. Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα καλά τους λόγια για την επικοδομητική τους ε, συνεργασία και έχουν παρατηρήσει δύο-τρία πράγματα. Αλλά θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω. Του και κάποιε άλλη επιτροπής που έχουν την, την κυρίω αρμοδιότητα, διότι εδώ έχουμε κάποια ευρύτερα ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει και τα ζητήματα εκείνα τα χειρίζονται οι συνάδελφοι εκείνη τη κυρίω αρμόδια ε, της Επιτροπής. Καλά τα λέει ο ότι είναι θέμα ε, και μεγαλύτερων επιχειρήσεων και όχι με μία ε, Εμείς πάντως βλέπουμε τα πράγματα από πλευράς ε, όχι τόσο ατομικών ελευθεριών όσο από πλευράς ε, επιχειρήσεων. Οπότε αυτό θα να πω για στον κύριο Χρόουτε, ότι συμφωνώ μαζί του. Προβληματιζόμαστε και όσον αφορά την προστασία του ιδιωτικού βίου και όσον αφορά τα κοινωνικά δίκτυα. Με μεγάλη μου χαρά ε, άκουσα ευτυχώς αυτά που μου είπαν ε, τα παιδιά μου να μην μπω στο facebook άκουσα και τι είπε η κυρία Νίμπλερ και αυτή που βοήθησε όσον αφορά το θέμα της privacy by design και θεωρώ ότι θα πρέπει ακριβώς να προσπαθήσουμε να πετύχουμε την επιδιωκόμενη ισορροπία. Ευθύνη, κατορισμός της ευθύνης όσον αφορά τη χρήση των δεδομένων, αλλά να μην βαρύνουμε υπερβολικά τον κόσμο με τυπικές υποχρεώσεις. Για να δούμε επομένω στη συνέχεια προθεσμίες και χρονοδιάγραμμα. Πρόεδρος. Ναι, 13 Ιουνίου. Απριλίου. Απριλίου. 12 η ώρα προθεσμοί για τροπολογίε. Για όσου θέλουν να καταθέσουν. Αν δεν θέλει να πει κανεί τίποτα άλλο, τελειώνουμε με αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη και το ρολόι μα λέει πώ έχουμε μισή ωρίτσα, αλλά δεν έχουμε άλλα σημεία στη ημερήσια διάταξη. Οπότε, καλή σα όρεξη. Το μπούστι.